Αγαπητοί συνάδελφοι, εφόσον είστε εδώ για την πρώτη στρογγυλή τράπεζα, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, λοιπόν, πάρτε θέσεις. Εάν δεν συμμετέχετε στην πρώτη στρογγυλή τράπεζα, παρακαλώ ε, να μεταβείτε στην άλλη αίθουσα. Κυρίε και κύριοι, ένα θερμό καλωσόρισμα σε αυτή τη στρογγυλή τραπέζα που θα εξετάσει το θέμα του ασύλου και τη μετανάστευση. Ε, εγώ είμαι επικεφαλής της Επιτροπής ε, Δημοσίων Ελευθεριών, Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιοσύνη. Ε, έχουμε μια μεγάλη, ένα μεγάλο κατάλογο μιλητών. Ε, σας υπόσχομαι ότι θα είμαι πολύ αυστηρό με το χρόνο έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν αλλά να γίνει ταυτόχρονα και μια καλή συζήτηση στην οποία θα συμμετέχουν όλοι. Τόσο ο γύρο τραπέζι μεταδίδεται στο διαδίκτυο, υπάρχει web streaming και καταγράφονται όλες οι ομιλίες. Υπάρχει διερμηνία σε μια σειρά από γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. Μπορείτε και να μιλήσετε και να ακούσετε ελληνικά. Αυτές είναι λοιπόν οι γλώσσες που μπορείτε, ε, μπορείτε να εκφραστείτε θα ήθελα να σα ενημερώσω επίση ότι ο, η Ισογγελή Τράπεζα για την σταθερότητα και την ευημερία στις χώρε, χώρες ε, λαμβάνει χώρα σε μια άλλη αίθουσα στην 3C50, ε, δεν πρόκειται να σας κουράσω με μια μακροσκελή εισαγωγή. Ήθελα μόνο να σας πω ότι η ιδέα αυτού του γύρω τραπέζης είναι να εξασφαλίσουμε ότι είναι να εξασφαλίσουμε ότι η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει θα μπορέσει να, να φτάσει σε όλους. Ε, θα πρέπει όντως ε, να ανέβει λίγο και το air εδώ, ο κλιματισμός, διότι κάνει ζέστη στην αίθουσα. Για να μπορέσει να λειτουργήσει ε, όλο αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θα μιλήσει μόλις 5 λεπτά ε, ο, ο Επίτροπος, καλωσορίζω και τον ε, Υπουργό, χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ μαζί μας, Υπουργός από την Ελλάδα, Πέντε λεπτά λοιπόν ο καθένα, ο επίτροπο και ο Υπουργό, ε, για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Είναι πολλοί εδώ ε, έμπειροι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα θέματα μετανάστευση. Χωρί λοιπόν να μακρηγορήσω στην εισαγωγή μου, να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον σε αυτό το γύρο τραπέζι μέσω και το web streaming, ε, ε μέσω της, των αναφορών που θα προκύψουν των εκθέσεων, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Έχουμε έναν αριθμό ρεκόρ νομοθετικών προτάσεων ε, στον τομέα του ασύλου. Ε, έχουμε πολύ έντονη δραστηριότητα. Θα αναφερθεί σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίω ο Υπουργό αλλά και τα διάφορα μέλη εδώ θα αναφερθούν ε, και στην πολύ έντονη δραστηριότητα όχι μόνο στην Ιταλία και στην Ελλάδα, στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά στο σύνολο τη Ένωση. Α προσπαθήσουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά και να μιλήσουμε και για λύσει. Λοιπόν, ο Επίτροπο Αβραμόπουλο πρώτα. Επίτροπος Έχετε πέντε λεπτά. Ε, πείτε μας πώς βλέπετε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, εάν κάτι έχει καταστήσει σαφές τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ότι χρειαζόμαστε όχι απλά μια ευρωπαϊκή αλλά μια παγκόσμια προσέγγιση για το θέμα της μετανάστευσης. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι πώς η μετανάστευση ε, μπορεί να ε, αποτραπεί ή να τη σταματήσουμε. Είναι πώς θα τη διαχειριστούμε. Η δυνατότητά μας ως Ένωση να ανταποκριθούμε θα καθορίσει το, την ίδια την Ένωσή μας, Τα αμυγός εθνικά μέτρα δεν αρκούν. Μας το έδειξε η κρίση. Δεν αρκούν σε επίπεδο κράτους μέλους, αλλά ούτε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη Ευρώπη για να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια, ένα πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα που να αντέχει στο μέλλον σε ό,τι αφορά το άσυλο. Θα πρέπει να εξαρθρώσουμε ε, και να κυνηγήσουμε τα κυκλώματα διακινητών. Θα πρέπει αυτοί που δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Ένωση να επιστρέψουν στις χώρες τους. Θα πρέπει να αυξήσουμε τέλος τις ασφαλές διόδους. Όμως, περισσότερη Ευρώπη δεν σημαίνει ότι θα αφαιρέσουμε αρμοδιότητες από τα κράτη-μέλη, όπως φοβούνται κάποιοι. Περισσότερη Ευρώπη σημαίνει μια καλύτερη και πιο κοινή διαχείριση μιας, απέναντι σε μια κοινή πρόκληση. Χρειάζεται μεγαλύτερη αλληλεγγύη και περισσότερη κατανομή ευθυνών. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός της μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Πέρα, παρά τις πολλές προσπάσεις που γίνουν στο παρελθόν, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα εθνικά συστήματα ασύλου. Αυτή ακριβώς η διαφορά είναι που οδηγεί ε, στις δευτερογενείς μετακινήσεις και στην αναζήτηση του καλύτερου τόπου ασύλου. Και βεβαίως αυτό ε, μεταθέτει τις ευθύνες μεταξύ κρατών μελών. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα αναρμονισμένο, ισχυρό και δίκαιο σύστημα ασύλου. Ένα σύστημα που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην ισότιμη κατανομή ευθυνών. Όπου καμία χώρα δεν πρόκειται να φεθεί να αντιμετωπίσει τέτοιες προκλήσεις μόνη τη. αλλά και ένα σύστημα το οποίο θα αντέχει στην κρίση. Εάν θέλουμε να κλείσουμε τα κενά, θα πρέπει τα εθνικά συστήματα ασύλου να ευθυγραμμιστούν με φιλόδοξο τρόπο, σεβόμενοι βεβαίως τι ευρωπαϊκές προδιαγραφέ και τις ευρωπαϊκές αξίες. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα του συστήματο, αλλά και για να εγγυηθούμε ισότιμη και αξιοπρεπή μεταχείριση των ετούντων άσυλο ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιτυχία όμως αυτής της μεταρρύθμισης τελικά εξαρτάται από την αλληλεγγύη. Η γεωγραφία ε, δεν μπορεί να καθορίζει την ευθύνη, η γεωγραφική θέση του καθένα. Το Δουβλίνο, όπως το γνωρίζουμε, απέδειξε ότι δεν αντέχει το τεστ του χρόνου και της εξέλιξης. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο Δουβλίνο, πιο δίκαιο, όπου η κατανομή των ευθυνών θα αποτελεί μέρος του συστήματος. Χρειαζόμαστε ε, ένα καλύτερο Δουβλίνο και αυτό πάει πέρα από το Δουβλίνο. Εάν θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη χωρίς εσωτερικά σύνορα, τότε χρειαζόμαστε μια προβλέψιμη και αποτελεσματική συμφωνία ε, σε ό,τι αφορά το σύστημα του Δουβλίνου. Λαμβάνω χώρα διαπραγματεύσει από το κρατομελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, υποστηρίζει το εγχείρημα για ένα τέτοιο μηχανισμό. Βεβαίω χρειαζόμαστε τη δέσμευση όλων των κρατών μελών, η οποία πρέπει να μεταφραστεί σε πολύ συγκεκριμένους και δεσμευτικούς νομικούς κανόνες. Ο σκοπός μας επίσης είναι να, να εξετάσουμε το θέμα των παράτυπων μετακινήσεων και να εξασφαλίσουμε ασφαλές οδούς εισόδου. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ε, επανεισδοχή, έτσι ώστε να υπάρξουν αυτές οι οδοί ασφαλείς και νόμιμες για όσους χρειάζονται και χρήζουν διεθνούς προστασίας. Χρειαζόμαστε επίσης ισχυρά εξωτερικά σύνορα για να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του Σέγγεν. Όπως γνωρίζετε την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισαν 32 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το, ο χώρος Σέγγεν. Πρέπει να διαφυλάξουμε ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Χαίρομαι λοιπόν που χάρη και στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε πλέον συστηματικούς ελέγχους στις βάσεις δεδομένων για όλους, όλους περνούν από τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Μαζί με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή, όλα αυτά έχουν ενισχύσει την ασφάλεια στα σύνορά μας. Πάνω από 1.600 εξωματικοί υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη ε, και τις χώρες εχμής και έτσι τα ευρωπαϊκά σύνορα προστατεύονται καλύτερα από ποτέ η εξωτερική και η εσωτερική διάσταση της διαχείρισης της μετανάστευσης συνδέονται άρρηκτα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ενισχύσει τις ρυπνεύσεις μας απέναντι στις τρίτες χώρες κλειδιά έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση στη ρίζα της στις χώρες προέλευσης, στις χώρες διαμετοκάμεσης, να αντιμετωπίσουμε τη διακίνηση, να βελτιώσουμε τις επιστροφές και να ενισχύσουμε τις νόμιμες οδούς. Δεν θέλουμε μια Ευρώπη οχυρό. Θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ανοιχτή και ανεκτική, αλλά και ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμίσουμε καλύτερα και την νόμιμη μετανάστευση και την κινητικότητα, όχι μόνο για αυτούς που χρειάζονται προστασία. Η πρόταση μεταρρύθμισης της μπλε κάρτας είναι μέρος αυτής της προσπάθειας. Θέλουμε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους μετανάστες με προσόντα, με δεξιότητες, διότι θα τους χρειαστούμε. Από την άλλη, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την παράτυπη μετανάστευση. Πρέπει να βελτιώσουμε την επιστροφή αυτών που δεν έχουν το δικαίωμα παραμονής. Η νέα εντολή της Ευρωπαϊκής Συνοριαφυλακής ε, θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Τα κράτη-μέλη όμως θα πρέπει να εφαρμόσουν και καλύτερα τους υπάρχοντες κανόνες. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της ένταξης. Διότι τελικά όλα όσα συζητάμε εδώ αφορούν την συνοχή των κοινωνιών μας στο μέλλον. Αφορούν το πώς μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Και γνωρίζουμε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι όλο και πιο ποικιλόμορφε. Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε ούτε από κοινωνικής ούτε από οικονομικής πλευράς. Μόνο μια επιτυχής ένταξη των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας επιτρέψει η μετανάστευση να αποτελέσει πραγματικά ευκαιρία και για αυτούς, αλλά και για το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας. Σε ένα πραγματικό πνεύμα αλληλεγγύης, εξαρτάται από όλους μας, η μετανάστευση να αποτελέσει ένα ευρωπαϊκό success story, διότι αφορά το μέλλον του συνόλου της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much, Commissioner. A few days ago... Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Πριν από λίγες μέρες, η Επιτροπή ε, Λίμπε και μια αντιπροσωπεία της επισκέφτηκαν την Ελλάδα. Είναι μια δύσκολη στιγμή. με λυπή χρηματοδότηση έχετε βρεθεί στην πρώτη γραμμή αντιμετώπιση της μετανάστευσης από την πρώτη στιγμή. Και γι' αυτό ο κύριο Μουζάλα, ο υπουργό που είναι υπεύθυνο για τα θέματα αυτά από την Ελληνική Δημοκρατία, θα μα μιλήσει για 5-6 λεπτά. Σα παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ε, Κλοντ, ε, σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το Ευρωκοινοβούλιο για αυτή την εκδήλωση και για την πρόσκληση που μου έκανε ε, είναι δύσκολο. Ε, θα ξεκινήσω, το έχω πει και άλλες φορές, ξαφνιαστήκαμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα. Η Ελλάδα με έναν φοβερά αδύνατο διοικητικό μηχανισμό και με μια πλήρη απειρία στην αντιμετώπιση των προσφύγων και μεταναστών. Βρεθήκαμε απροετοίμαστοι σαν χώρα, βρεθήκαμε απροετοίμαστοι σαν Ευρώπη. Ο Γιουνκέρο, πρόεδρος, εγκαίρος έδωσε το σύνθημα του Resettlement Relocation Returns η Ευρώπη δεν μπόρεσε να το εφαρμόσει, ε, αντιμαχίες, διαμάχες, δυσκολίες. Γιατί ξαφνιαστήκαμε. 20 χρόνια γίνεται πόλεμος. Από το Αφγανιστάν μέχρι τη Λιβύη. Νομίζω ότι συμμετοχή είχαμε και ευρωπαϊκά κράτη σε αυτό. Γιατί λέμε με τόση αθωότητα ξαφνιαστήκαμε. Πώς θα γίνει να μην επιτρέψουμε να ξαναξαφνιαστούμε γνωρίζοντας ότι ο πόλεμος δεν μπορεί παρά να έχει τέτοια αποτελέσματα και αποφεύγοντας τον πόλεμο. Πώς μπορούμε να μην ξαναξαφνιαστούμε γνωρίζοντας ότι οι κλιματικές αλλαγές, το ξέρουμε από τώρα, η φτώχεια, η διαφθορά, η πείνα οδηγεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε μετανάστευση και σε προσφυγιά. Τα γεγονότα 2015 μέχρι τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκία ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες τράνζιτ από την Ελλάδα δέκα μέρες χρόνος παραμονής. Διαχειριστήκαμε αυτή τη κρίση με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως στην αρχή με την τεράστια αλληλεγγύη του λαού μας και αλληλεγγύη λαών οργανώσεων από ξένα κράτη. Δεν επιτρέψαμε να αναπτυχθούν ακραία ρατσιστικά, ξενοφοβικά φαινόμενα. Είναι προσκρίση το πόσο καλά τα καταφέραμε, που κάναμε λάθη, κάναμε λάθη, δεν γίνεται να μην κάνεις λάθη, δεν έχει όμως αυτή η συζήτηση σήμερα αυτό εδώ το νόημα. Κλείνει η οδός των Δυτικών Βαλκανίων παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι ροές από 5.000 την ημέρα πέφτουν στις 2.500 την ημέρα. Εγκλωβίζονται 60.000 άνθρωποι που αντιστοιχεί με 560.000 ανθρώπους στη Γερμανία. Δημιουργούνται δομένοι πριν την ειδωμένη ο Πειραιάς, το ελληνικό. Ξεκινάμε έναν απίστευτο αγώνα. Δημιουργούμε μέσα σε λίγους μήνες 50.000 θέσεις φιλοξενίας. Είχαμε χίλιες. Οι 50.000 θέσεις φιλοξενίας δεν είναι καλές. Επιτρέπουν όμως να διαλύσουμε την ιδωμένη τον Πειραιά και τώρα πια στο τέλος και το ελληνικό. Και να τις κάνουμε κάθε μέρα και καλύτερες. Αποκτούμε μια εμπειρία στη διαχείριση και στην υποδοχή των προσφύγων και μεταναστών που η χώρα μου δεν την είχε. Με τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας οι ροές αποκτούν έναν χαρακτήρα ελέγξη. Η κατάσταση στην ενδοχώρα βελτιώνεται. Οι προσπάθειες που κάναμε για αυτά ήταν τεράστιες. Σας είπα και πριν, όταν ξεκινήσαμε χίλιες θέσεις, 50.000 θέσεις, ε, πέντε μήνες ε, μετά την διάλυση της ειδωμένης. Ε, Άσυλο, το ιδρύσαμε το 2013. Με 200 άτομα ξεκίνησε το άσυλο, μας έπιασε η κρίση. 800 άτομα σήμερα. Έχουμε καλό χρόνο έκδοσης ασύλου και προσφυγών σε σχέση με το τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ΕΑΣΟ μπορεί να μαρτυρήσει γι' αυτό. Ε, και είμαστε η δεύτερη χώρα σε αριθμό αιτήσεων ασύλου υγεία εμβολιασμούς κάναμε από την ειδωμένη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα παιδιά έχουν ξεκινήσει πάνε σχολείο, αλλάζουμε τη τροφή με κάσ, αντί συσίτια, βελτιώνουμε τις κατοικίες από τα κακά κάμπ, περνάμε στα καλά κάμπ και στα αξιοπρεπή κάμπ και στη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών ετούντων άσυλο στα διαμερίσματα. Για τα ασυνόδευτα έχουμε ξεκινήσει με 280 θέσεις, έχουμε αυτή τη στιγμή 1.400 και 200 safe zone και βέβαια για κάθε βελτίωση που σας λέω ένα καινούριο κύμα θα την καταργήσει. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι το Σεπτέμβριο δεν θα έχουμε κανένα ασυνόδευτο έξω από δομή. Εάν μέχρι το Σεπτέμβριο έρθουν άλλα 700 ασυνόδευτα θα διαψευστώ. Θέλω με αυτό να πω ότι η δράση μας στην διαχείριση της μετανάστευσης εξαρτάται από ένα παράγοντα απρόβλεπτο που πρέπει να μπορούμε να τον προβλέψουμε. Τη ροή. Σε όλη αυτή την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση μας βοήθησε. Μας βοήθησε. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Με πολύ μεγάλες δυσκολίες στη συνεργασία μας. Οι θεσμικές οργανώσεις μας βοήθησαν μας βοήθησαν με πολύ μεγάλες δυσκολίες στη συνεργασία μας. Δεν μοιραστήκαμε το πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πει μοιράζομαι. Μας βοήθησαν με ΕΑΣΟ, μας βοήθησαν με Frontex. Είναι εδώ, δουλέψαν υπέροχα. Δεν μοιραστήκανε το πρόβλημα. Και φτάνουμε στο σημείο σήμερα όπου με κυρώσεις θα γίνει η αλληλεγγύη, χρειάζεται, αλλά δεν είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε όταν κυρώσεις επιφέρουν την αλληλεγγύη. Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω μια εμπειρία και για να μην ξαναξαπνιαστούμε. Οι προηγούμενοι ομιλητές μιλήσανε και δικαίως μονάχα για τον δρόμο Αφρική-Λιβύη-Ιταλία. Αυτό προϋποθέτει ότι ο δρόμος Ασία-Τουρκία, ε, κοντινή Αφρική, Αιγαίο, ε, Ελλάδα και από εκεί πάλι η Ευρώπη δεν πέφτει. Η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας ισχύει. Ξέρω ότι για τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες φωνές. Δεν την χαρακτηρίζω καλή, κακή, οτιδήποτε. Λέω, είναι μια πολύ χρήσιμη συμφωνία. Εάν έχει ελαττώματα, εάν έχει ελαττώματα και έχει ελαττώματα, εάν έχει γκριζε ζώνες και έχει γκριζε ζώνες, να διορθωθούν εκεί που δημιουργούνται. Διότι κοιτάξτε να δείτε, από 21 Τρίτου του 16 που έγινε η Συμφωνία Ευρώπης Τουρκίας μέχρι 21 Δευτέρου του 17 26.940 αφήξεις. Από 24 Τετάρτου του 15 έως 20 Τρίτου του 16 977.700 αφήξεις. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρώ ότι είναι μια ευκολία, αλλά ενέχει και μια υποκρισία. Το να ξεκινάμε να αντιμετωπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη στιγμή που πατάνε το πόδι του στην Ευρώπη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ξεκινάνε από τη στιγμή που φεύγουν από το Αφγανιστάν, που φεύγουν από την Ιγυρία, που φεύγουν από το Σουδάν, που τους σκοτώνουν στη Συρία από εκεί. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει εκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους αυτούς, πρόσφυγες και μετανάστες, να τους δώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα που δικαιούνται και την πρόσβαση στο άσυλο πριν μπουν στη βάρκα. Μέσα σε processing center υπό την ευθύνη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με όλα αυτά που προβλέπει η συνθήκη της Γενέβη και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Με processing center μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε θα αφήσουμε τους ανθρώπους στο τρίτο μεγαλύτερο εμπόριο, παράνομο εμπόριο, το εμπόριο των σμάγκλων. 500.000 διασώσεις έχουμε κάνει στη θάλασσα. Η Ιταλία κάνει τα αντίστοιχα. Πριν μπουν στη βάρκα, πριν μπουν στη βάρκα οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε ασφαλείς διαδρόμους για τους πρόσφυγες. Νόμιμους δρόμους μετανάστευσης. Η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας ισχυρίζομαι μπορεί με βελτιώσεις, μπορεί με παρεμβάσεις να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω λέγοντας το εξής. Και στο καινούριο Δουβλίνο η Ευρώπη βοηθάει τις χώρες υποδοχής. Δεν μοιράζεται. Και επειδή δεν μοιράζεται και το καινούριο Δουβλίνο θα καταπέσει όπως έπεσε το πρώτο σε οποιαδήποτε μεγάλη κρίση. Γνωρίζω την βαθιά δουλειά που έχει γίνει εδώ πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο για το κοινό άσυλο και για το σύστημα Δουβλίνου και πόσο πολύ έχει κουραστεί και η κυρία Βίξτρον. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Είσαστε η άμεση επαφή της Ευρώπης με τους λαούς της και χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε να παντρευτούν οι δύο αυτές τάσεις και η βοήθεια που δίνεται στις χώρες πρώτης υποδοχής να συνδυαστεί με το μοιράζομαι ιδάλλως πάλι θα καταπέσει. Στη συνεργασία μας είχαμε πολλά προβλήματα. Με την Ευρώπη, με την Επιτροπή, με τις θεσμικές οργανώσεις, μαθαίναμε. Και εμείς και η Ευρώπη. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στη συνεργασία μας ήταν προβλήματα που λυνόντουσαν. Ήταν προβλήματα που μάθαμε να τα λύνουμε και ευτυχώς και ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Τηλιανίδης ε, και ο Γιούνκερ και πάρα πολλοί κόσμος μας βοήθησε σε αυτό το πράγμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε και λύνουμε τα προβλήματα με υποχωρήσεις μας, με κατανόηση καλύτερη. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν θα μπορούσαμε να λύσουμε. Το να μην υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόριο οφθαλμού εάν θέλουμε να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ και μπορεί να προσέξατε ότι και ο Επιτροπός και ο Υπουργός μίλησαν λίγο παραπάνω. Δεν έχω ακόμα βρει την τόλμη και το θάρρο που χρειάζεται για να σα διακόπτω, αλλά πλησιάζουμε, γιατί έχουμε 39 ομιλητέ. Θα τα καταφέρουμε και θα τα βγάλουμε πέρα. Έχω βρει με τι τρόπο αυτό το πετύχω. Πολύ απλά. Όλοι μπορούν να μιλήσουν μέχρι 4 λεπτά. Αν θέλετε χρησιμοποιήστε και λιγότερο, 2 λεπτά. Αν μιλήσετε 2 4 λεπτά, 4 κατά το όριο. Στα 4 λεπτά πολύ απλά θα σα διακόπτω και θα περάσουμε στον επόμενο σα. Το υπόσχομαι θα το κάνω μεταξύ των 39 ατόμων αυτών είναι και άτομα τα οποία έχουν, όπως είπε ο υπουργό εργαστεί ακούραστα για θέματα μετανάστευσης στο παρελθόν, στα θέματα της, του Δουβλίνου, σε θέματα επανεγκατάστασης, να ακούσουμε την άποψή σας και έχουμε και προσκεκλημένους από διάφορες χώρες που πλήττονται από την κρίση. Ας ε, περάσουμε λοιπόν κατευθείαν στους ομιλητές μας. Θα αναφέρω τους τρεις επόμενους. Κύριε Μέτσολα, Σλάιν και Σεσίλια Βίξτρομ. Θα ξεκινήσουμε με την Ρομπέρτα Μετσόλα. Εδώ είναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ξεκινήστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η διάσταση της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε είναι πραγματικά σχεδόν απίστευτη. Εξακολουθεί ο κόσμος να χάνει τη ζωή του στις θάλασσές μας. Εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και ω πολιτικοί έχουμε καθήκον να τοποθετηθούμε και να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι στατιστικά στοιχεία χωρί όνομα. Αν ένα πράγμα έμαθα τα τελευταία χρόνια που ήμουν μέλο του Κοινοβουλίου είναι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε γρήγορη λύση και μαγική ε, ασημένια σφαίρα, αν θέλετε, για την επίλυση των προβλημάτων. Θα πρέπει να σκεφτούμε και να έχουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχουν ε, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με καταπήγουσε λύσει. Θα πρέπει να υπάρχει ένα βιώσιμο σχέδιο και θα πρέπει να υπάρχουν ε, ευρωπαϊκέ υπηρεσίε όπω η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Άσυλο και να έχουν σε πόρου και προσωπικό για να τα βγάζουν πέρα. Η αλληλεγγύη θα πρέπει να αποτελεί την αρχή επί τη οποία θα βασίζεται οποιαδήποτε δράση για τη μετανάστευση και οποιαδήποτε τέτοια δράση θα πρέπει να περιλαμβάνει και μέτρα που θα στοχεύουν τα εγκληματικά κυκλώματα Παράλληλα, θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ αυτών που χρήζουν ε, προστασίες και αυτών που έρχονται στην Ευρώπη για δουλειά. Και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι άνθρωποι που φεύγουν από τον πόλεμο έχουν δικαίωμα προστασίας, όντω αληθεύει ότι αυτό δεν ισχύει σε μετανάστευση για όλου. ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την εργασιακή μετανάστευση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ελέγχουν την αγορά εργασία του και αυτά τα κράτη-μέλη και η Ένωση θα πρέπει να φροντίσουν να καλύψουν τα, χάσματα, τα ενδεχόμενα χάσματα στην αγορά σε θέματα επανεκατάσταση των ε, ατομών που χρήζουν διεθνού προστασία. Θα πρέπει επιτέλου, λοιπόν να καταστούμε μια ένωση κοινών αρχών και ευθυνών. Θα πρέπει να υπάρξουν και νόμιμοι διόδοι και καλύτερη προσέγγιση στην επανεγκατάσταση. Γιατί αν το πετύχουμε αυτό, τότε ο κόσμο δεν θα ε, αισθάνονται υποχρεωμένο να μπαίνει σε σαπιο κάραβα και να χάνει τη ζωή του στη θάλασσα. Σε θέματα ασφάλεια δεν μπορούμε να στρωθοκαμιλίζουμε. Σε θέματα ασφάλειας υπάρχει ανησυχία και φόβη μεταξύ των πολιτών μα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκπληρώνουν τις ευθύνε του στα εξωτερικά σύνορα αν θέλουμε να απαλληλθούν αυτές οι ανησυχίε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ακραίους και τους λαϊκιστές να κατέχουν αυτή την ιστορία και αυτό λοιπόν θα πρέπει να ενισχύσουμε παράλληλα και τα εξωτερικά σύνορα. Ξέρουμε ότι δεν ε, δικαιούται προστασία όποιο, όλοι όσοι καταφτάνουν στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτού που δεν ε, χρήσουν προστασία σε το Δουβλίνο. Η νομοθετική διαδικασία που βρίσκεται να εξελίξει θα πρέπει να γίνει σεβαστή και θα πρέπει να έχουμε χρόνο στα πλαίσια του Κοινοβουλίου να χαράξουμε το μελλοντικό δρόμο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα άτομα για την επικράτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση για την ενσωμάτωση και θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια Θα πρέπει φυσικά να δώσουμε ευκαιρίες, αλλά πρέπει να ακολουθούν τις αξίες μας ε, όλοι όσοι εντάσσονται στην κοινωνία μας. Θα πρέπει να δούμε τα αίτια και να κατανοήσουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη δέσμευση για να επιλύσουμε τη γεωπολιτική κατάσταση και τα γεωπολιτικά προβλήματα της εποχής μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και την εξωτερική διάσταση του θέματος. Η Ευρώπη θα πρέπει να βοηθήσει να αναπτυχθούν δυνατότητες στα τρίτα κράτη που τελικά θα δημιουργήσουν ε, συνθήκες ασφαλέστερες ε, σε κράτη πιο κοντά στις πατρίδες του κόσμου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, πάντα ηγέτης παροχή βοήθειας προς την Αφρική. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε και επενδύσεις. Ένα Marshall Plan για την Αφρική. Κύριε Πρόεδρε, αν ένα μήνυμα θα κρατήσουμε από σήμερα είναι το εξή. Δεν μπορούμε να χάσουμε την ευαισθησία μα στο γεγονό ότι η μετανάστευση είναι ανθρώπινο ζήτημα. Είναι αληθινοί άνθρωποι με αληθινέ ζωέ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για όλο τον κόσμο σε τέτοια ζητήματα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ρομπέρτα. Ε, καλό θα ήταν να συστηνόμαστε όλοι γιατί για τους προσκεκλημένους μας ε, είναι σημαντικό. Ε, η Ρόπερτα Ματσούλα είναι βουλευτής του ΕΛΚ και ήταν εισηγητρία για μια ρεαλιστική προσέγγιση στη μετανάστευση. Επόμενη ομιλήτρια θα ήταν η Σεσίλ Κιέγκε, η άλλη συνεισηγήτρια για το ίδιο θέμα, όμως δεν μπορούσε να παραβρίσκεται. Οπότε τη δική της χρονοθυρίδα παίρνει η Έλλη Σλάινεν από την ομάδα των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και θα μιλήσει εκ μέρους της Εσίλ Κιέγκε, ε, η κυρία Σλάιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί χρόνια, έξι από τα 28 κράτη-μέλη παλεύουν μόνα τους με τις αιτήσει ασύλου που υποφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερώτηση είναι λοιπόν, είναι αυτό αλληλεγγύη και ίση κατανομή ευθυνών ε, τις οποίες απαιτούν οι συνθήκες στο άρθρο 78 και 80 όχι. Το περασμένο Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, η πρώτη σύνοδο στο ΙΕ για του πρόσφυγε και του μετανάστε διοργανώθηκε, διότι 86% όλων των εκτοπισμένων παγκοσμίω ε, είναι ε, στα χέρια των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι αρχηγοί κατά δύο κυβερνήσεων ε, δεσμεύτηκαν για δικαιότερη κατανομή ευθυνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώ υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μα θα αναλάβει το δικό τη μερίδιο ευθύνη, αλλά οι πολιτικέ τη Ένωση συγκαλύπτουν και όπως ε, τώρα μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, αναθέσουν εξωτερικό τη διαχείριση των συνόρων μας όπως η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ε, η Συμφωνία με τη Λιβύη, όλες οι, όλοι οι κατάλογοι περιθεωρήσεων και οι κατάλογοι ασφαλών χωρών. Όλε οι συμφωνίε από το Συμβουλίο είναι όνειρο. Είναι απαράδεκτο κυβερνήσει που θα έπρεπε να σέβονται τι δεσμεύσει του ω προ την μετεγκατάσταση σε 1,5 χρόνο να έχουν μετεγκαταστήσει μόνο 20.000 ανθρώπου ενώ ο Καναδάς σε τέσσερις μήνες κατάφερε να κατακαταστήσει 40.000. Δεν είναι θέμα αριθμών ημέσων το ζητούμενο, αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης και των εθνικών εγωισμών. Είναι μια πρόκληση που κανένα κράτος μελό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του. Πρέπει να υπάρξει μια κατάσταση και μια λύση βιώσιμη για όλους. Όπως ε, τόσες ε, ιστορίες από την Ιταλία μας δείχνει, ε, υποδοχή των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο είναι ευεργετική για τι ίδιε τι τοπικέ κοινότητε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια λύση ευρωπαϊκή σε μια σφαιρική προσέγγιση και να έχουμε την ε, ε, πρόκληση των ε, Ευρωπαίων που να αντιμετωπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι κοινέ ευθύνε θα πρέπει να κατανέμονται δικαίως. Η δάλο είναι παιδιάστικη η αντίδραση. Θα πρέπει μακροπρόθεσμα να βεβαιωθούμε ότι ξεπερνάμε την υποκρισία του συστήματος του Δουβλίνου και όπως ζήτησε τον περασμένο Απρίλιο το Δουβλίνο να πάμε σε κεντρική ανάληψη των ευθυνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό θα ε, προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το κριτήριο των ε, παράνομων εισόδων και να υπάρχει ε, το κριτήριο του ε, κράτους μέλους διαμονής για να δούμε τους ε, νόμιμους δεσμούς που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Στην Ιταλία, στα σύνορα ε, Ιταλίας Ελβετίας είδαμε χιλιάδες άνθρωποι να κοιμούνται στους δρόμους ε, κοντά στη λίμνη του Κόμου. Εδώ θα πρέπει οι άνθρωποι αντί να κοιμούνται στους δρόμους ε, να δούμε γιατί είναι θύματα ενός συστήματος που τους αφήνει δύο χρόνια να περιμένουν την οικογενειακή επανένωση. Χρειαζόμαστε περισσότερους νομικούς, ε, νόμιμους δρόμους για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών δεν μπορεί μόνο όσοι προσπαθούν να αποφύγουν τον πόλεμο, ε, μάλλον ε, όσοι προσπαθούν να αποφύγουν τον πόλεμο, να μην μπορούν να βοηθηθούν εδώ. Θα πρέπει να δούμε και άλλα θέματα, όπω η οικονομική μετανάστευση ή η διαφυγή από τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει να ε, έχουμε διαχείριση των συνόρων στην Αφρική και να ε, δώσουμε ευκαιρίες στους νέους Αφρικανούς. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε την ακτοφυλακή της Λιβύης. Να μην ε, ακούμε ιστορίες ότι πυροβολούνται μετανάστες από την Ιταλική ακτοφυλακή. Θα πρέπει να φροντίσουμε για τη συνέπεια των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ξένες πολιτιστικές Πολιτικέ ε, για τι εξωτερικέ υποθέσει, δημοσιονομικέ πολιτικέ, οικονομικέ πολιτικέ. Στα πλαίσια τη ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνάδελφοι, αυτό που προσπαθούμε να σα πούμε είναι ότι χρειάζεται όχι απλώ ένα αποτελεσματικό σύστημα ασύλου ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εδώ παίζεται ολόκληρο το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρέπει να δείξουμε στου πολίτε γιατί χρειάζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αντιμετωπίσουμε τι κοινέ προκλήσει με κοινέ λύσει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Υπουργό προηγουμένω αναφέρθηκε στο έργο τη Σεσίλια Βέξτρομ, που είναι ευρωβουλευτή από την Άλντε και είναι και εισηγητή, πιο σημαντικό, για την αναθεώρηση τη ε, συνθήκη του Δουβλίνου. Κυρία Σεσίλια Βέξτρομ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορούμε και δεν θα πρέπει ποτέ να είμαστε αφελείς για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η υπηρεός μας σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, αλλά εκ παραλλήλου δεν μπορούμε και ποτέ δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον φόβο και το λαϊκισμό να υπαγορεύσουν τις αντιδράσεις μας σε όλα αυτά. Στο ζενήθ του, της μεταναστικής κρίσης το 2015 περίπου μετανάστες αυτές στι ακτέ στις ακτές μας. 1,3 ετούντες άσυλο σε μια ήπειρο 500 εκατομμύριων ε, ανθρώπων. Δεν είναι ούτε καν το 1,3% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τότε λοιπόν είχαμε μοιραστεί δίκαια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τις ευθύνε μας, αυτό θα είχε σημαίνει, θα σήμαινε ότι μια πόλη 10.000 κατοίκων θα είχε λάβει επιπλέον 30 άτομα. Λίγες οικογένειες. Τόσο πια αντίνατον θα ήταν αυτό. Το 2015 αποτύχαμε, αποτύχαμε γιατί η πολιτική ασύλου είχε βασικά λάθη και χάσματα, γιατί δεν μοιραστήκαμε τις ευθύνες με τέτοιο τρόπο και αποτύχαμε γιατί δεν υπήρξε αλληλεγγύη καθόλου μεταξύ κρατών μελών το τρέχον σύστημα του Δουβλίνου οδηγεί σε χάο και ουσιαστικά αποτελεί πόλο έλξη για αυτού που ξέρουν ότι στην πράξη θα μπορέσουν να επιλέξουν όποιο κράτος μέλος θέλουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και έχει προκληθεί μια πραγματικά παράλογη κατάσταση, όπου κάθε κράτος μέλος έχει συμφέρον να μην καταχωρήσει κανέναν από τους έτοντες άσυλο, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα ήταν υπεύθυνο το κράτος μέλος για την αξιολόγηση και τη διεκπαιρέωση της αίτησής τους. Εννοείται ότι ούτε έλεγχος ασφάλειας θα υπάρχει αν ο κόσμος δεν καταχωρίζεται. Οι καλές ειδήσει, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι είναι δυνατόν να υπάρξει διαφορετική πολιτική. Μία πολιτική, ένα σύστημα με καλή διαχείριση, όπου κάθε κράτος μέλος θα αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τους έτοιμπες άσυλο. Αυτό θα μας επέτρεπε να κάνουμε σωστό έλεγχο ασφάλειας για όλους όσοι καταφθάνουν. Θα μας δώσει έλεγχο και πάλι για την κατάσταση και θα εξασφαλίσει στους ετούντες άσυλο ότι θα είναι δίκαιη η εξέταση της αίτησής τους. Ανεξάρτητα από το ποιο κράτος μέλος τελικά θα αξιολογήσει την αίτησή τους, ένα τέτοιο σύστημα δίκαιο για το άσυλο δεν σημαίνει ότι μπορεί να μείνουν όλοι, αλλά ότι όσοι πληρούν τους όρους για διεθνή προστασία θα μπορέσουν να παραμείνουν και όσοι δεν πληρούν τους όρους θα επιστραφούν με γρήγορα αλλά και αξιοπρεπή τρόπο. Όλοι οι πολιτικές, Όλες οι πολιτικές μάχες των τελευταίων χρόνων, όλα τα ad hoc μέτρα τα οποία αναγκαστήκαμε να πάρουμε και ο αγώνας ε, για προς τα κάτω των κρατών μελών για τους όρους υποδοχής είναι τα αποτελέσματα, οι συνέπειες της έλλειψης ενός σωστού συστήματος για το άσυλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την πραγματευτική ομάδα της οποίου ηγούμε ως εισηγήτρια για τον κανονισμό του Δουβλίνου θα είναι επικοδομητικό σε όλες τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, Ωστόσο, θα υπενθυμίσουμε στα κράτη-μέλη ότι η αλληλεγγύη στο τομέα του ασύλου αποτελεί βασική αρχή, η οποία κατοχυρώνεται και στι συνθήκε. Και ω εκ τούτου, δεν αποτελεί κάτι το προαιρετικό. Ποτέ. Σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχτούμε αποδυνάμωση και συμβιβασμού μόνο και το συμβιβασμό. Γιατί το μέλλον τη ε, Υπήρου εξαρτάται από την κοινή ανάληψη των ευθυνών μα και γιατί οι πολίτε περιμένουν πραγματικά να πετύχουμε αποτελέσματα και να φτιάξουμε αυτό το σύστημα το οποίο έχει προβλήματα. Κάποιος είπε ότι πάνω απ' όλα θα πρέπει να υπάρχει ελπίδα. Θέλω να προσθέσω ότι αυτή που θα πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Σεσίλια. Πολύ ενδιαφέρουσες τις τρεις πολύ δυνατές. Ο Χωσέ Καρέρα τώρα από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου και ο κύριος Ντεμπρουκέρ, ο ερευνητής του Κέντρου έρευνα. Ε, για δύο λεπτά παρακαλώ Ευχαριστώ πολύ. Συνήθως ε, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και επί τόπου, οπότε και εδώ θα κινηθώ γρήγορα, αλλά πρέπει να έχει νόημα παρέμβαση. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, θα ήθελα να πω κάτι που είπε και ο κύριος Γιούνκερ ε, ε, και η κυρία Μογκερίνη. Ε, όλοι οι υπουργοί αναγνώρισαν ότι έχουν γίνει πολλά. Και όλοι είπαν ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Και οι τρεις ευρωβουλευτές σε, σε κάποιο βαθμό από διαφορετικά πρίσματα αυτό το κοινό μήνυμα μας έδωσαν. Εγώ θυμάμαι τον Απρίλιο του 2015 τα πρώτα δέκα σημεία δράσης του Συμβουλίου και λίγο μετά υπήρχε μια ατζέντα για την ε, μετανάστευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αργότερα το ίδιο έτος ε, βεβαίως ε, εμφανίστηκε η έννοια του hot spot. Είχαμε την πρώτη σύνοδο κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια έως το, το, το, το του 2016 φτάσουμε στη συμφωνία και τη δήλωση με την Τουρκία. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε και κάποιες νέες προτάσεις, μετά είχαμε τη σύνοδο κορυφή της Βαλέτας και βεβαίω όλα τα σχέδια δράσης, τα συμπεράσματα. Αυτό που έχουμε δει λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια απάντηση, μια ευρωπαϊκή απάντηση, εντατική, με τρεις βασικούς πυλώνες ο πρώτος πυλώνας έχει να κάνει με, ένα μηχανισμό κρίσης, ένα μηχανισμό απάντησης στην κρίση. Νομίζω εδώ μιλάνε μόνα τους τα αποτελέσματα. Μπορεί να υπάρχουν βεβαίως ε, ε, αφιλεγόμενα στοιχεία, αλλά έχουμε πετύχει αδιαμασβήτη πρόοδο. Από την άλλη έχουμε τον πυλώνα που αφορά την ομοθετική ε, τροποποίηση που είναι εξελίξη και υπάρχει και ο τρίτος πυλώνας η εξωτερική διάσταση, η μετανάστευση σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Μου έχουν μένει λεπτά βέβαια, αλλά να πω ότι και στου τρει του πυλώνες η Άσο ήταν παρούσα. Είμαστε ένα σημαντικός παράγοντας και στην απάντηση και στη διαχείριση. Είμαστε στο επίκεντρο πολλών νομοθετημάτων ε, που συζητούνται αυτή τη στιγμή και που θα εγκριθούν, ελπίζουμε, και επίσης ε, εξετάζουμε, αντιμετωπίζουμε και τη ρίζα ε, της μετανάστευσης, της ρίζες της μετανάστευσης. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Μωράης, ε, λέει ο κύριος Ντεμπρούκερ, θα είμαι σύντομος. Ε, είμαι νομικός σε ένα δίκτυο που έχουν φτιάξει συνάδελφοι από όλα τα κράτη-μέλη, να σας πω ποια είναι η άποψή μας ε, για το ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Η δική μας ε, ανάλυση είναι ότι η κρίση την οποία ε, ζούμε δεν είναι μια κρίση προσφύγων. Είναι μια θεσμική κρίση, είναι μια κρίση θεσμών. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει και αλλάζουν οι αρχές της. Κανονικά οι ευρωπαϊκές πολιτικές ε, ναι είστε στο C250 και κάθεστε κύριε Λεμπρίκερ έχεις να σας πιάσουν η κάμερα γι' αυτό λέω τον, τον που κάθεστε το 250 κάθεστε μάλιστα συνεχίστε παρακαλώ Περνάμε λοιπόν από την ε, εφαρμογή πολιτικών από τα κράτη-μέλη σε μια κοινή εφαρμογή δηλαδή με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε σε αυτή τη μετάβαση και δεν βλέπουμε φως, διότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα τούνελ. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα λοιπόν είναι αλληλεγγύη. Χρησιμοποιείται συχνά αυτή η λέξη, αλλά πρέπει να πω ότι δεν νομίζω να έχουμε ξεκινήσει ε, σε μια σωστή βάση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μιλάει για ασφάλεια για αλληλεγγύη μάλλον και ευθύνη. Και αυτές οι δύο έννοιες τις αντιπαραθέτει. αν, αν δει κανεί τι λέει το άρθρο 18 της συνθήκης, έχουμε την αρχή της αλληλεγγύης και, και της κοινή κατανομής ευθυνών. Δεν είναι αντιτιθέμενες έννοιες. Ε, και κανείς δεν έχει καταλάβει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπέρασμα της Πρατισλάβα αλλά και αλλού, δεν μιλάει για fair sharing, δεν μιλάει για ισότιμη κατανομή ευθυνών, μιλάει για αλληλεγγύη έναντι της ευθύνης. Ενώ πρέπει, πρέπει να μιλάμε για αλληλεγγύη η οποία ενισχύεται από μια ισότιμη κατανομή ευθυνών. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε στα κείμενα των συνθήκων εδώ. Okay, our next three speakers will... Ε, ο ομιλητές είναι η Χέλγα Στίβενς και ο τρίτος είναι ο Δημήτρης Δημητρίου. Αρχίζουμε με τη Χέλγα Στίβενς από την ομάδα ECR για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Λέει ο πρόεδρος πριν ξεκινήσετε, η Χέλγα Στίβενς, Φεράρα και Μάρτιν. Μάρτιν Κλίντ. Ζητώ συγγνώμη. Η κυρία Χέλγα Στίβενς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα στον γύρο τραπέζι αυτών μαζί σα και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να, ακούμε, να ακούσουμε την άποψή σα για την επιστροφή της ε, διαδικασία τη επιταχυνισμένη και την ε, ενσωμάτωση. Και είναι σημαντικό το ότι βρίσκονται εδώ όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 40 ομιλητές ε, έχουν καταγραφεί και θα είναι ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων. Κυρίε και κύριοι, πιστεύω ότι θα πρέπει να φυλάξουμε τα σύνορά μα και για να έχουμε και πάλι έλεγχο θέλουμε να, υπάρχουν, να υπάρχει υποστήριξη στην κοινωνία μα για την υποδοχή πραγματικών ε, προσφύγων. Πέραν αυτού, για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. πριν από κάποια χρόνια έγιναν κάποιες ε, σύλληψεις και έτσι ξεκίνησε μια αμφισβήτηση. Αλλά για να βάλουμε ένα τέλος ε, στο χάος ε, στην Ελλάδα, στα σύνορα με την Ελλάδα και με την Ιταλία, αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια συμφωνία με την Τουρκία. Είναι λοιπόν απαραίτητη, με επιτακτική ανάγκη να βρούμε τρόπο να ελέγχουμε τα σύνορά μας. Οι μετανάστευσες αποστέλλονται επιστρέφονται σε ασφαλείς χώρες, λέει η αρχή της ε, μη Μιλάμε όμως και για ασφαλείς λιμένες. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο οι μετανάστες ε, να επιστρέφονται, να μεταφέρονται στην Ιταλία μετά την διάσωσή τους ή μήπως ε, αρκεί και κάτι άλλο τώρα, για παράδειγμα, μεταφέρονται συστηματικά στην Ευρώπη για, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και έτσι λοιπόν ουσιαστικά ευνοούμε τους διακινητές. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δόγμα του δικαιώματος για άσυλο στη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Helga. Συγγνώμη που σας διάκοψα πριν. Η Λόρα Φεράρα είναι συντονίστρια και εισηγήτρια για θέματα διαδικασιών χορήγησης ασύλου. Δύο λεπτά. Νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να μιλήσουμε για θέληση και όχι λύσεις, γιατί οι λύσεις συμπίπτουν με τη θέληση όταν υπάρχει. Δηλαδή δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε στις συζητήσεις για τους ετούντες άσυλο. Θα πρέπει να είναι μια συζήτηση που να σχετίζεται μια γενικότερη θέληση διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών ολιστικά ή να δούμε κατά πόσο θα χειραγωγούμε αυτό το φαινόμενο όπως έγινε μέχρι τώρα από όλα τα κράτη-μέλη. Χειραγώγηση για πολιτικούς λόγους και εν εκλογών. Επειδή θέλουμε να χειραγωγήσουμε το εκλογικό σώμα. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να δούμε κατά πόσο θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτή την προοπτική ή να προβάλλουμε μια ολιστική πολιτική για να επιλύσουμε το θέμα των μεταναστευτικών ε, ροών ε, ολιστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ απευθύνομαι στα κράτη-μέλη, γιατί τα κράτη-μέλη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αύριο θα συνεδριάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο δυστυχώς εκπροσωπεί εθνικούς εγωισμούς. Μιλάμε για λύσεις σήμερα, αλλά τις λύσεις τις έχουμε ήδη. Μιλήσαμε για 160.000 μετανάστες που θα πρέπει να μετεγκατασταθούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουν, ε, έχει γίνει επανεγκατάσταση μόνο 12.000 και 16 αντιστοίχως από την Ελλάδα και την Ιταλία. Και ε, δυστυχώς ε, υφίστανται την κατάσταση λίγα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φαίνεται ότι θέλουν πολύ να εξουδετερώσουν αυτή την αναθεώρηση για να μην υπάρχει κατανομή ετούντων άσυλο σε όλα τα κράτη-μέλη. Ως προς την αναθεώρηση της Frontex, ο πρόεδρος Γιούγκερ μας μίλησε για την ακτοφυλακή σαν ένα μεγάλο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μας στην Ιταλία μας είπαν ότι δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Δεν είμαστε σε θέση. Ε, δυστυχώς η Ιταλία είναι ε, μια χερσόνησος που βρέχεται από τρεις πλευρές και συμπεριλαμβάνει και δύο άλλα μεγάλα νησιά. Κρίμα λοιπόν που δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλη την ε, ακτογραμμή. Ε, λυπάμαι, μου είχε υποθεί ότι έχω τέσσερα λεπτά. Έχουμε 180.000 ελεύσεις, 150.000 από τις αρχές ε, του 2015 και του 2016. Ως προς την συμφωνία με την Τουρκία, αυτό είναι ένας άλλος στόχος ε, με την Ευρωπαϊκή, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι όμως μακρόπνοη λύση. Έπειτα είναι λύση για ποιον. Για την οδό των Βαλκανίων, σίγουρα δεν είναι λύση για την οδό της Μεσογείου. Επίσης, μιλάμε για 58 ε, εκατομμύρια, τα οποία αφορούν ε, αναλήψη υποχρεώσεων από μία μόνο χώρα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ξενοφοβία και τον ρατσισμό καθώς και το λαϊκισμό. Θα πρέπει να τηρήσουμε τις συνθήκες. Μιλάμε για το άρθρο 80 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνει λόγο για αλληλεγγύη μεταξύ όλων κρατών μελών. Θα πρέπει να τηρούμε τις συνθήκες στο δινεκές. Διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αδύναμη στους ισχυρούς και ισχυρή στους αδύναμους. Ευχαριστώ, Λόρα. Ίσως σας είχαν δοθεί τέσσερα λεπτά αρχικά, αλλά τώρα συνάδελφοι θα πρέπει να αρκεστείτε στα δύο. Και λυπάμαι αν είχατε αυτή την ένδειξη. Μάρτιν Κλούς είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων από το Σλοβακικό Κοινοβούλιο και από την ομάδα ECR. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Στη Σλοβακία λέμε ότι εκεί που τελειώνει η επικοινωνία αρχίζει η σύγκρουση. Γι' αυτό χαίρομαι για την σύγκληση αυτής της διάσκεψης. Η χώρα μου δεν έχει δεχτεί τις θεσμευτικές ποσοστώσεις εδώ και αρκετό καιρό γιατί από την πείρα μας έχουμε διαπιστώσει ότι η χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όταν ήταν αλληλέγγυες δυστυχώς δεν ε, είχαν μία αντίστοιχη πορεία και από τις άλλες χώρες. Είχαμε δεχτεί πολλούς μετανάστες από το Ιράκ που είτε επέστρεψαν στο Ιράκ είτε μεταφέρθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ίδιο έχουν τονίσει και η Τσεχία και η Λετωνία. Οι πρόσφυγες ε, δεν είναι σακιά με πατάτες που μπορούμε να μεταφέρουμε κατά από μία χώρα στην άλλη. Κατά τη Σλοβακική Προεδρία μιλήσαμε για ευέλικτη αλληλεγγύη, δηλαδή αλληλεγγύη μέσα στα πλαίσια του εφικτού από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Θεωρούμε ότι η αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου, σύμφωνα με την οποία εμείς θα πρέπει να δεχτούμε μετανάστες ή να υποστούμε κυρώσεις, δείχνει ότι θα υπάρχει και μία ανωδική τάση των ναζιστικών και λαϊκιστικών δυνάμεων στις χώρες μας. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα επί της ουσίας. Φυσικά θα πρέπει να προωθήσουμε την νόμιμη μετανάστευση από νόμιμε, νόμιμους διάβλους και από την Τουρκία και από τη Λιβύη. Έχουμε το παράδειγμα της Αυστραλίας και άλλων χωρών που έχουν υπεράκτιες, υπεράκτιους καταβλισμούς και ίσως αυτό αποθαρρύνει τη διακίνηση των μεταναστών για λόγους κέρδους αποκλειστικά. Επίσης, έχουμε αποσύρει την υποχρέωση θεώρηση στη Γεωργία και Ουκρανία ως μια χειρονομία καλής θέλησης προς αυτές τις χώρες. Και αυτό είναι ένα θετικό παράδειγμα της μετανάστευσης ε, επί της ουσίας. Δημήτρης Δημητρίου ο κύριος Καμίνης και Μισελ Λεβόη που είναι ο κύριος Δημητρίου, ε, είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών ποθέσεων από την Κυπριακή Βουλή. Λία έχουν πληγεί περισσότερο από αυτή τη μεταναστευτική κρίση, σε αυτό πιστεύω συμφωνούμε οι πλήστοι εδώ πέρα και συμφωνούμε το εφιστάμενο πλαίσιο χρειάζεται αναθεώρηση. Η ευθύνη και η αλληλεγγύη όλων των κρατών μελών προ όλα τα κράτη-μέλη χρειάζεται να είναι δεδομένη και αφορά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γεωγραφία είναι ο μόνος παράγοντας σε αυτή όλη την εξίσωση που δεν μπορεί να αλλάξει. Ένα αποτελεσματικό λοιπόν σύστημα ασύλου δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς αυτοματοποιημένο, υποχρεωτικό και δίκαιο μηχανισμό ανακατανομής των δικαιούχων. Η διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο συστηματικής παρακολούθησης με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Η ενίσχυση των εξωτερικών σύνορων με την αποτελεσματική παρακολούθηση από την σύνοριοφυλακή είναι δε σημαντική και απαραίτητη. Οι αυξητικές τάσεις της διαθαλάσσης αφήξεων στην Κύπρο από την Τουρκία υποδεικνύουν ενδεχόμενη δημιουργία νέας παράτυπης μεταστευτικής οδού, γεγονός που απαιτεί την επαγρύπνηση όλων των εμπλεκομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία και ως μία πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση συνολικά, με χειροπιαστά αποτελέσματα, στρατηγική στόχευση για το μέλλον, με αξιοποίηση της τεχνολογίας και μείωση της γραφειοκρατίας. Τα αποτελέσματα αυτά θα είναι πιο άμεσα και πιο πιστικά προς τις πραγματικές προθέσεις και την πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ και τώρα ο Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηνών, για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Αθήνα, όπως ξέρετε, έχει πληγεί από τις ροές των προσφύγων. Δεν είχαμε πρώτερη εμπειρία αντιμετώπισης ε, ροών προσφύγων τέτοιας κλίμακας, όμως ε, ήμασταν οι πρώτοι που αντιδράσαμε όταν ε, η κρίση αυτή εκδηλώθηκε το καλοκαίρι του 2015. Ήταν καθήκον μας να συνεισφέρουμε για να βρεθούν λύσεις, να δώσουμε ένα παράδειγμα ως πρωτεύουσα της Ελλάδας για τη διαχείριση των μεταναστών. Δεν είχαμε πόρους, δεν είχαμε αρμοδιότητες, δεν υπήρχε εθνική στρατηγική αρχικά. Ήταν όμως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν θέμα αξιοπρέπεια αλλά και κοινωνική συνοχή. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να δώσουμε ένα χώρο δημοτικό ε, για τα πρώτα κέντρα ε, επεξεργασία. Κάναμε δομικέ αλλαγέ στο Δήμο και δημιουργήσαμε ένα κέντρο συντονισμού όπου συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οργανώσεις της πόλης όμως ε, οι πολίτες και γενικότερα οι τοπικές αρχές ανά την Ευρώπη έχουν ε, ένα πολύ σημαντικό ρόλο απέναντι στο το φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε στις κοινότητές τους. Ε, είχαμε την πρωτοβουλία αλληλέγγυων πόλεων με την υποστήριξη του Eurocities Network το ξεκίνησε η Αθήνα αυτό. Οι πόλεις είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους πρόσφυγες και να βοηθήσουν με την ε, διαδικασία μετακίνησής τους και στέγασής τους είχαμε σημαντικά, σημαντικά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε δύσκολα αναγνωρίστηκαν ε, αυτά βέβαια και με τα πλαίσια της αστικής ατζέντα, της urban agenda πέρυσι πρέπει να υπάρχει άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση όμως να υπάρχουν περισσότερες αρμοδιότητες για τους Δήμους και να υπάρχει καλύτερο συντονισμός με τις άλλες, τα άλλα επίπεδα διακυβέρνησης. Στην Αθήνα οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είναι αποκλεισμένοι εδώ και μήνες ε, και είναι, βρίσκονται σε μια κατάσταση αδιεξόδου που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι πολλές διαφορές. Ε, οι διαφορές από τις πόλεις, από τις χώρες στις οποίες έρχονται. Εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Υπάρχει αυροσκεπτικισμός. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η μετανάστευση είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, um, Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Και τώρα ο Μισελ Λεβόη από μια μη κυβερνητική οργάνωση που έχει βάσει στις Βρυξέλλες. Ε, ναι, θα ήθελα να επαναπροσανατολίσω ε, λίγο τη συζήτηση. Εδώ στο 496 είμαι. Στο 496 να μιλήσω λοιπόν για τους μετανάστες, διότι νομίζω ότι επικεντρωθήκαμε πολύ στο σύστημα ασύλου. Ε, και βεβαίως ε, είναι πολύ οι φάκελοι που εξετάζει το Κοινοβούλιο γύρω από το άσυλο, αλλά ε, δεν υπάρχει 100% ποσοστό ε, χορήγησης ασύλου, ούτε 100% επιστροφών. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί και θα υπάρχουν και πολλοί παράνομοι παράτυποι μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν συστήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ. Τέσσερα σύντομα σημεία. Πρώτα απ' όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζονται και για τους μετανάστες που δεν έχουν χαρτιά. Δεν είναι κάτι που είναι υποδιαπραγμάτευση. Το, λέει, το λένε τα Ηνωμένα Έθνη στις προδιαγραφές τους. Για να συμβεί αυτό στην πράξη πρέπει να έχουμε δικλείδες ασφαλείας. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρχουν πάροχοι ε, υπηρεσιών ε, που δεν θα κάνουν τη δουλειά τους. Θα πρέπει ε, ε μέσω ενδεχομένω της οδηγίας για τα θύματα ε, εγκλημάτων ε, ότι υπάρχει περίθαλψη για οποιονδήποτε, οποιοδήποτε θύμα ε, εγκλήματος. Ε, πώς θα γίνει το πραγματικότητα. Ίσως να μην πρέπει ε, ε οι ε, άνθρωποι χωρίς χαρτιά να υπόκεινται σε διακρίσεις. Θα πρέπει αυτό να αφορά και την οικογενειακή επανεισδοχή αλλά και την εργασία. Την οικογενειακή επανένωση, αλλά και την εργασία. Αυτό αφορά και άλλους τομείς οικονομικούς, όχι μόνο την δηλωμένη εργασία. Το τρίτο ζήτημα είναι τα παιδιά. Τα παιδιά μπορούν ακόμα να είναι υποκράτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι υπάρχει συνένεση σε επίπεδο δικαιωμάτων ότι αυτό δεν είναι προ συμφέρον του, ότι είναι παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού. Πώ μπορούμε να βρούμε λοιπόν εναλλακτικέ στην κράτηση, ε, πώ μπορούμε να έχουμε διαδικασίε διαχείριση εξατομικευμένη, ώστε και τα παιδιά και οι οικογένειέ του σιγά σιγά να βγουν από το καθεστώ κράτηση ε, και να έχουν ε, πρόσβαση σε μια εξωπρεπή κατοικία. Και βεβαίω ε, οι συνθήκε εργασία. είναι σημαντικό να ισχύουν για όλου του εργαζόμενου. όποιο και να είναι το καθεστώς διαμονή του. Υπάρχει νομοθεσία ευρωπαϊκή, η οποία όμω έχει περίπλοκου μηχανισμού σε ό,τι φορά τι δυνατότητε, για έναν μετανάστη χωρί χατιά να εργαστεί. Ε, δεν είναι όμω ε, για την ώρα δυνατό οι άνθρωποι αυτοί να προσφύγουν όταν παραβιάζονται τα δημοσιογραφικά του δικαιώματα. Πώ θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα αυτό. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε ε, νομοθετικές ε, διασυνδέσει εδώ, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη, ε, links μάλλον που θα θα σας στείλω για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το όλο αυτό εγχείρημα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Μισελ. Οι τρει επόμενοι ομιλητέ τώρα είναι η Μάρλεν Μπιόρκ, Τζοάν Γκούντι και Βιντσέντζο Μελόνι. Ξεκινάμε με τον Μάλεν Μπιόρκ που είναι η συγγήτρια από την ομάδα Γκούε έχει τέσσερα λεπτά στη διάθεσή τη. Έτσι λέει εδώ. Ε, δεν είναι δικό μου το χαρτί, τέσσερα λεπτά λέει εδώ. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Τόντι, θα ήθελα ο τίτλος του πάνελ αυτού να είναι προστασία των προσφύγων και να δημιουργείται ένα σύστημα υποδοχή που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό διακυβεύεται. Αυτό είναι που δεν επιτυγχάνουμε. Για μένα και πολλού από του συναδέλφου μου εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, η γενική κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη μετανάστευση και του ασύλου δεν είναι εντάξει. Διότι ε, επικεντρώνεται στο να κρατήσει απ' έξω του ανθρώπου. Το ακούσαμε και σε αυτή την αίθουσα. Στι χώρε μα γίνεται ένα αγώνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά των εξτρεμιστικών δυνάμεων και τη ξενοφοβία. Κάποιοι θέλουν να κάνουν την ήπειρό μα, τι χώρε μα, ε, να την μετατρέπουν σε μια ισοστρεφή, περίκλειστη ζώνη. Δεν θέλουμε να ε, υποκύψουμε στι κοσμοθεωρίε του και τι πολιτικέ του, ούτε έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα. Το αντίθετο. Εμεί έχουμε την ευθύνη να παράσχουμε εναλλακτικέ λύσει και απόψει. Πρέπει να δημιουργήσουμε τι ανοιχτέ κοινωνίε στι οποίε θέλουμε να ζούμε. Και έχουμε όλοι μεγάλη ευθύνη να το κάνουμε αυτό. Επίσης αυτό σημαίνει, και θα μιλήσω και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο και σε κάποιου από του συναδέλφου, ε, θα στραφώ προς αυτούς λέγοντάς τα αυτά, πρέπει η αλληλεγγύη προ του πρόσφυγε να ε, επανέλθει μεταξύ των προϊόντων μας ε, και στην χάραξη πολιτικών και στην ατζέντα μας. Δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ω θηρευτέ ασύλου ως ε, εκμεταλλευτές αυτούς που ετούνται άσυλο. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται εδώ γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Συνάδελφοι, πρέπει να έχουμε ασφαλής διόδους προς την Ευρώπη. Ο μόνος τρόπος να σταματήσει η λαθρεμπορία ανθρώπων είναι να δημιουργηθούν ασφαλείς οδοί. Και πολλοί έχουν κάνει έκκληση, αλλά πολλές λίγες πρωτοβουλίες έχουμε δει στην πράξη. Έχουμε μόνο ε, έναν ε, μια προσπάθεια μετακατάσταση που είναι η μόνη λύση προ την δημιουργία νόμιμων οδών για την νόμιμη μεταμετανάστευση. Είναι η μόνη πολιτική επιλογή και η μόνη συγκεκριμένη λύση για πολλού ανθρώπου. Χρειάζονται περισσότερε νόμιμε οδοί. Πέρα από τη μετακατάσταση θα θέλαμε να δούμε και τι ανθρωπιστικέ θεωρήσει, τα ανθρωπιστικά προγράμματα υποδοχή και την ε, ε, γρήγορη και σύντομη οικογενειακή επανένωση. Αλλά για να επανέλθω στην ε, μετεγκατάσταση. Πρέπει να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει ένα εργαλείο ε, για να ε, ελεγχθεί η μετανάστευση, να επιβληθούν συμφωνίες επανεισδοχής ή να ε, υποθούνται η ελεύθερη κυκλοφορία των μεταναστών. Είναι ένα αρχιτεκτόνιμο από το και κάποιε χώρε εδώ και δεκαετίε. Είναι ένα εργαλείο διεθνού αλληλεγγύη που αντιμετωπίζει συγκεκριμένε ατομικέ ανάγκε διαβίωση για συγκεκριμένου ανθρώπου. Έτσι θα πρέπει να την ακλάβουμε τη μετακατάσταση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη λοιπόν να εντείνουν τι προσπάθειέ του και η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει έναν μείζονα ρόλο στην ετατικοποίηση αυτή. Συνάδελφοι, πρέπει να πούμε όχι και στην εξωτερική, ε, ε, την εξωτερική τη ευθύνη για τα σύνορα. Ε, καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στην Τουρκία, την Λιβύη, την, την, η οδός ε, Τουρκίας-Ελλάδας, ε, ουδέποτε ξανά είχαμε ουδεποτε ξανεχαμε νεκρούς στην Μεσόγειο. Το ότι δεν βλέπουμε του νεκρούς δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι ασφαλεί, ε, φίλοι μου. Επίση, οι παραστατευτικέ ομάδε στη Λιβύη δρούν ως ε, αυτεπάγγελτε εκτοφυλακέ για να σταματήσουν του λαθρομετανάστε. Αυτό δεν σώζει κανέναν, ίσα ίσα απειλεί τι ζωέ πολλών ανθρώπων. Ε, Απευθυνόμενοι λοιπόν στο Συμβούλιο να πω ότι πρέπει να τα πάτε καλύτερα. Πρέπει να δημιουργήσετε μια συμμαχία που να ε, φέρει αποτελέσματα. Δεν μπορείτε να αθρίζεστε στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Όσου θέλουν να κλείσουν τι πόρτε τη Ευρώπη έχουν τη λιγότερη βούληση. Πρέπει να σεβαστείτε τι διεθνεί υποχρεώσει, το, το διεθνέ δίκαιο και να βρείτε λύσει που να προσφέρουν βιώσιμε ευρωπαϊκέ απαντήσει προστατεύοντα του πρόσφυγε και μετανάστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μάλιν. Και τώρα ο Γενικός επισμηναγός της ακτοφυλακής για τρία λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις επιχειρησιακές, διότι από τις, ε, από τις παρεμβάσεις που έγιναν είδα ότι υπάρχουν πολλά που μπορούν να υποθούν. Βάσει των ε, συμβάσεων που διέπουν ε, τις δραστηριότητε διάσωσης, είναι σαφές ότι κάθε χώρα έχει ένα συγκεκριμένο τομέα ευθύνης, ε, ε, περιοχή ΣΑΡ όπως ονομάζεται. Τώρα τι συμβαίνει στη Μεσόγειο. Συμβαίνουν τα εξής. Στην πράξη η Λιβύη και η Τινησία έχουν δεχτεί τη σύμβαση του Αμβούργου, αλλά ουδέποτε δήλωσαν ποιο είναι ο χώρος, η περιοχή Σάρ που τους αναλογεί. Κατά συνέπεια, χιλιάδες χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα θάλασσας μεταξύ του νότιου ε, ορίου της Μάλτας για τις διασώσεις και την περιοχή της Λιβύης αλλά και την ακτή της Λιβύης και της Τινησίας δεν φυλάσσονται από κανέναν. Δεν είναι διοργανωμένες και κανείς δεν έχει την ευθύνη για τη διάσωση εκεί. Πρόκειται για μια τεράστια μαύρη τρύπα όπως θα έλεγα. Ε, τι λένε οι συμβάσεις. Οι συμβάσεις λένε ότι η χώρα που λαμβάνει μια κλίση για διάσωση πρέπει να δράσει, ε, να παρέμβει. Ακόμη και αν η κλίση προς βοήθεια είναι εκτός της περιοχής ευθύνης της. Ε, κατά συνέπεια ε, όλα αυτά είναι γνωστά στις εγκληματικές οργανώσεις και βεβαίως αυτές οι οργανώσεις φροντίζουν να εξοπλίσουν τα σκάφη, σκάφη τα οποία είναι αυτοσχέδια και ιδιαίτερα φορτωμένα με γυναίκες και παιδιά που πρέπει να πω εν παρενθέσει ότι από τις αρχές ε, του 2017 ως σήμερα είναι 70.000 αυτοί που διασώσαμε, των οποίων 10.000 ασυνόδευτα παιδιά. Κατά συνέπεια λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι κλήσεις για βοήθεια από τις ίδιες εγκληματικές οργανώσεις πηγαίνουν προς την Ιταλική ακτοφυλακή. Πηγαίνω στο επιχειρησιακό κέντρο τη Ιταλική ακτοφυλακή. Ε, ε, του νόμου λοιπόν πρέπει να παρέμβουμε. Αν δεν το κάνουμε και γίνει κάτι, κάτι πάει στραβά, μια τραγωδία, ένα ναυάγιο, τι συνέπειε, τι ποινικέ τι έχει η Ιταλική ακτοφυλακή, αν θέλουμε να το δούμε από αυτή την οπτική γωνία. Από τη δική μα οπτική γωνία, βέβαια, προέχει ηθική επιταγή να παρέμβουμε. Οπότε, εάν δεν υπάρξει παρέμβαση, σίγουρα θα υπάρξουν νεκροί. Γι' αυτό λοιπόν η Ιταλική εκτοφυλακή, το Όντι, ε, καλείται να διαχειριστεί, να διοργανώσει επιχειρήσεις διάσωσης στην Μεσόγειο, στη μισή Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο, να μην ξεχνάμε ότι έχουν παράλληλα 23 χώρες. Κι όμως η Ιταλία βρίσκεται να διοργανώνει δραστηριότητες διάσωσης στη μισή Μεσόγειο, γιατί τις κλήσεις τις λαμβάνει η Ιταλία και πρέπει να παρέμβει. Και επειδή καμία χώρα δεν μπορεί να παρέμβει στη θέση της, διότι οι κλήσεις έχουν ε, να κάνουν με αυτή την περιοχή, τη μαύρη τρύπα που σας ανέφερα. Γι' αυτό το κύκλωμα είναι κλειστό. Και επειδή οι διαστηριότητε διάσωσης γίνονται από την Ιταλική εκτοφυλακή, από την Ιταλία, αυτοί που διασώζονται ε, μεταφέρονται στην Ιταλία. Αυτό, γι' αυτό ακριβώς πέρσι είχαμε 180.000 άτομα μετά τη διάσωση. Τη διάσωση. Και μετά τα γεγονότα της Αλβανίας, από το 1991 και μετά, η Ιταλική εκτοφυλακή συντώνησε επιχειρήσεις που έφεραν ε, διάσωση 90.000 ατόμων σε 26 χρόνια. Εκ των οποίων όμω, όπως έλεγα προηγουμένως, το μεγαλύτερο αριθμό στα τελευταία δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια του 2016 συντονίσαμε σε μία μόνο μέρα 53 επιχειρήσει διάσωση, βοήθεια και διάσωσης για 5.000 άτομα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό η εκτοφυλακή μόνη τη με τα δικά τη μέσα και μόνο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τα διάφορα συστήματα και μηχανισμοί που ε, λειτουργούν ε, στην περιοχή αυτή, η U4Med, ε, η Frontex, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει να συνεισφέρουν. Ευχαριστώ που σήμερα οι μη κυβερνητικέ οργανώσει έχουν έρθει ω εκεί. Διότι χάρη σε αυτέ τι οργανώσει, χάρη σε αυτέ τι εμπορικέ ε, παρουσίες έστω, καταφέρνουμε παρόλα αυτά να προσφέρουμε διάσ, επιχειρήσεις βοήθειας και διάσωσης. Τα εμπορικά σκάφη προσφέρουν βοήθεια. Το 2014 έπρεπε να μετατρέψουμε χίλια εμπορικά ε, και να τα καλέσουμε να ενισχύσουν τι προσπάθειε βοήθεια και διάσωση. Χάρη λοιπόν στις μη οργανώσει, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αυτά ε, είναι πλέον εφικτά. Ε, λυπούμε από χρόνο με τόσο λίγο, αλλά είχα πάτος τόσα πολλά να πω. Ε, σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Um, <clears throat> ε, ναι, και εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για όλους όσοι συμμετέχουν για τον τόσο λίγο χρόνο που έχουμε και επίσης πρέπει να εκφράσω την ευχαριστή, την ευχαριστή, ευχαριστίες μας προς όσους συμμετέχουν και προσπαθούν να βοηθήσουν σε αυτή την κρίση. Ο Τζάνι Γκούντι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για δύο λεπτά. Ή Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία να μιλήσω εκ μέρους του ΦΡΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Ο Οργανισμό ε, Θεμελιδών Δικαιωμάτων ασχολείται με τα θέματα μετανάστευση και ασύλου, ιδίω στο επίπεδο του δικαίου, προ τα ευρωπαϊκά ε, θεσμικά όργανα και προκειμένου να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Χάρτα των Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε του νομοθέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με την απαραίτητη έμπειρο γνωμοσύνη και πρόσφατα το πράξαμε αυτό σε μια σειρά από νομικέ νομοδοτήσει που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναδιατύπωση των προτάσεων που αναδιατυπώνουν την πρόταση Eurodac, καθώ και ε, τα όσα αφορούν τα κέντρα υποδοχή τη μετανάστευση. Σύντομα θα υπάρξει και μια γνωμοδότηση για το αίτιο. Κατά δεύτερον, η μετανάστευση και το άσυλο είναι, όπω γνωρίζετε, ένα χώρο υψηλή προτεραιότητα για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν μπορώ να το θέσω διαφορετικά, διότι το κοινωνικό κεκτημένο ε, εξελίσσεται ε, γοργά και είναι ύψη τη σημασία όχι μόνο να προσφέρουμε υπηρεσίε για την κάλυψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στι νέε προτάσει, αλλά να έχουμε πραγματικά και η μελέτη αντικτύπου για τα θεμελιώδη δικαιώματα με ένα εύρωστο ε, σύστημα και τις ανάλογες εγγυήσεις στα νομοθετικέ στις νομοθετικές μας προτάσεις. Κατά τρίτον, για να προστατευτούν τα παιδιά ε, στα πλαίσια της μετανάστευσης από την εκμετάλλευση, την βία και την ε, εμπορία, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται ότι το παιδί είναι παιδί και ω τέτοιο αντιμετωπίζεται. Τα παιδιά τη μετανάστευση δεν πρέπει να ε, πέφτουν αντικείμενο μεταχείριση ω μετανάστε, αλλά ω παιδιά. Ε, και θα πρέπει όσα προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού να ισχύουν για όλα τα παιδιά. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα παιδιά που ετούν άσυλο και τα παιδιά που μεταναστεύουν, ασχέτω από το που προέρχονται και χωρί καμία δικαιωτική μεταχείριση. Τέταρτον και τελευταίο, σε επιχειρησιακέ δραστηριότητε, η ΦΡΑ ε, προσφέρει συνδρομή στα hot spot στα κάτι και παρίσταται στα ελληνικά νησιά εδώ και ένα χρόνο. Ε, Επίση, ε, συστηματικά έχουμε επισκεφτεί τα hot spot τη Ιταλία, προσφέροντα εμπειρογνωμοσύνη για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, την ώρα που μιλάμε, έχουμε στείλει συνεργάτε μα στη Λέρο για να συνδράμουν του ευρωπαϊκού θεσμού, τι ελληνικέ αρχέ και άλλε φορεί στην αντιμετώπιση τη κατάσταση επιτόπου. Παρ' όλα αυτά, ε, βασική τομή προτεραιότητα είναι η αναθεώρηση του συστήματος για την κυδαιμονία, η πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση και η αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών και της εκμετάλλευσής τους. Θα σταματήσω εδώ και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πολλά θα μπορούσαν να λεχθούν, πολλά περισσότερα, αλλά σας ευχαριστώ που είσαστε πειθαρχημένοι και αναφέρεστε στα σημεία κλειδιά και μόνο. Αγαπητοί συνάδελφοι, έρθει είναι σχεδόν 5.30. Θα έπρεπε να λήξει η πρώτη αυτή συνεδρία. Δυστυχώς ο Επίτροπος πρέπει να αποχωρήσει και θα έπρεπε να έχει φύγει ήδη από τις 5, αλλά κατάφερε να μείνει μαζί μας λίγο περισσότερα. Εάν ύψαστε πειθαρχημένοι, θα κρατήσουμε το χρόνο μας. Ο κύριος Χάμπλ είναι ο πρόεδρος της Τσεχικής ε, Δημοκρατίας για θέματα που άπτουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Είμαι πεπισμένος ότι οι πολλοί μετανάστες οι οποίοι φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούν άσυλο απαρτίζονται από δύο βασικές ομάδες. Η πρώτη είναι οι πρόσφυγες ε, με βάση το διεθνές δίκαιο και μπορούν να τύχουν προστασίες, διεθνούς προστασίας, αλλά και μια μεγάλη ομάδα που δεν είναι πρόσφυγες, και που δεν έχουν παρά απειροελάχιστες ελπίδες προστασίας, αλλά και εκείνοι παραμένουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας σε δύο προτεραιότητες. Πρώτον, θα πρέπει να στυλιτεύσουμε αυτούς που οργανώνουν την μετακίνηση αυτών που δεν είναι πρόσφυγες η Frontex ε, μαζί με τις Αφρικανικές Μυστικές Υπηρεσίες εκπώνησαν μία έκθεση η οποία με ακρίβεια και καταλυπηρό τρόπο αποδεικνύει την ύπαρξη αυτών των δικτύων που μεταφέρουν ανθρώπους από την Αφρική που δεν είχαν καν πρόθεση να γίνουν μετανάστες, αλλά τους ε, πείθουν να διαπλέψουν τη Μεσόγειο. Και μετά είναι πολύ δύσκολο να παρέμβουμε στη Μεσόγειο. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δική μας νομοθεσία και ιδιαίτερα την νομοθεσία περιχορήγησης ασύλου. Όποιος ε, δεν λαμβάνει άσυλο τότε θα πρέπει να απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν γίνεται έμπρακτα. Και δυστυχώς οι κυβερνήσεις δεν ανταποκρίνονται. Θα ήθελα να παραμείνετε στα δύο λεπτά, σας παρακαλώ, έτσι ώστε όλοι να μιλήσουν. Θα δω επίσης πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί αρχίσαμε αργά με αυτή τη συνεδρία. Τώρα θα έπρεπε να αρχίσει η επόμενη. Υπό τον κύριο Δίας Μέρα, άρα θα μπορέσει κάποιος ίσως να με συμβουλέψει. Σας παρακαλώ να αρκεστείτε στα ε, δύο λεπτά. George Crowell από την Ιρλανδική Βουλή. Uh, chairman, I'm pleased θα χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα το απόγευμα για να συμμετέχω στη συζήτηση. Μου έκανα πάρα πολύ εντύπωση αυτά που άκουσα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του, μεταναστευτικού. Όπω ανέφεραν όμω και οι προηγούμενοι μελετέ, όλοι οι μετανάστε δεν είναι απαραίτητα και πρόσφυγε. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναζήτηση λοιπόν αλληλεγγύη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την τοποθέτηση των ε, μεταναστών και υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς μετανάστες. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζονται εργατικό δυναμικό και θέλουν να, θα έπρεπε να δίνουν βίζες για το προσωπικό, για τους ανθρώπους αυτούς. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά σε δύο λεπτά, αλλά θα πρέπει να, ε, να γίνεται μια κατηγοριοποίηση των μεταναστών. Ε, οι μετανάστες δεν είναι ε, που μπορούμε να τα αφήσουμε όπου να είναι και να περιμένουμε να βγάλουν πέρα μόνες τους. Θα πρέπει λοιπόν να, καταλάβουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καμία διάθεση να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται και φεύγουν ε, με την πρώτη ευκαιρία. Το σύστημα που έχουμε λοιπόν δεν είναι ικανοποιητικό σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Ούτε γι' αυτό έχουμε χρόνο να μιλήσουμε. Τελευταία δύο σημεία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την εγκληματικότητα που συνεπάγεται η μετανάστευση. Και τελευταίο σημείο, για να μην ξεπεράσω το χρόνο μου, είναι ότι θα πρέπει να φροντίσουμε και τους φτωχούς ε, πολίτες ε, που λάπτισαν τις χώρες ε, της Αφρικής και τώρα λαιλαπτούν το εργασιακό σύστημα. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι διακινητές, θα πρέπει να πληρώνουν για να μένει ο κόσμος, οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Εγώ είμαι από την Ιρλανδία. 17 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ε, είναι Ιρλανδοί. Είμαστε εμπειρογνώμονες, ειδικοί σε θέματα μετανάστευσης. Ευχαριστώ κύριε Πίτερ Μπόσμαν, δήμαρχος από την πόλη του Πυράν στην Σλοβενία. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και γι' αυτό θα μιλήσουμε και θα κάνουμε δύο σχόλια για τις πρακτικές με τις τρίτες χώρες. Η μετανάστευση ήταν η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατάρτισε ένα σχέδιο. το οποίο υποτίθεται ότι θα επέλυε κάποια από τα προβλήματα της μετανάστευσης, όπως τα αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη. Η μετανάστευση ήταν και θα είναι όσα τύχη και να αρθώσουμε, όσους φράχτες και οτιδήποτε άλλο και να αρθώσουμε, θα είναι ένα θέμα. Το πλαίσιο συνεργασία έχει λειτουργήσει υπό την έννοια ότι εντελώς βράχει πρόθεσμα μείωσε τον αριθμό των θανάτων. Δυστυχώς δεν τους έχει απαλείψει εντελώς. Λειτουργεί λοιπόν Ό,τι και αν λέμε για τη συμφωνία με την Τουρκία, κάτι πετύχαμε. Δυστυχώς, η οδός της Μεσογείου, και πρέπει να πω ότι η Ιταλία ήταν τα θέματα αυτά 5-6 χρόνια, αλλά υπήρχε και η οδός της Ιταλίας. Αυτή η οδός λοιπόν αποτελεί πρόβλημα. Το πρώτο τμήμα της ε, συμφωνίας ε, του πλαισίου συμφωνία λειτουργεί. Το δεύτερο τμήμα, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό, είναι η συνεργασία με τις χώρες της Αφρικής προκειμένου να ξεκινήσουν να αναπτύσσονται. Όχι να επιβληθούν ευρωπαϊκές λύσεις στην Αφρική, αλλά εταιρικέ σχέσεις. Κάποιος ανέφερε προηγουμένως το πόσο φθηνό είναι το εργατικό δυναμικό. για τις ομίλους στην Αφρική. Αληθεύει αυτό. Τέσσερα λεπτά. Όχι, όχι. Κάτι έγινε, κάποιο λάθος έγινε. Για να λειτουργήσει λοιπόν το πλαίσιο της εταιρικής σχέσης χρειάζονται αλληλεγγύη και τεράστιες επενδύσεις μακροπρόθεσμα. Και είναι το τελευταίο σημείο. κόσμος μιλάει για την ενσωμάτωση. Δεν σημαίνει παντού το ίδιο όμως. Σημαίνει ότι ζούμε σε μια κοινωνία με μεγάλη ποικιλία ως προς το πολιτισμικό υπόβαθρο και υπάρχει σεβασμό. Και νομίζω ότι ο κόσμος ε, περιμένει ότι οι μετανάστες που θα έρθουν θα είναι σαν αυτούς. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό και μετανάστες που πήγαν στην Αμερική. Ακόμα Ιρλανδοί αυτό που καλούνται. Αλλά είναι Αμερικανοί. Εγώ είμαι Αφρικανός. Επέλεξα να είμαι Σλοβαίνος και πιστεύω στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές αρχές. Thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σκάκελερ. Είναι Ευρωβουλευτή για τους πράσινου και εισηγήτρια τη έκθεση για τη μετεγκατάσταση. Αν θα μπορούσατε να μην μακρηγορήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ Κλοντ. Πολλοί από του αδέλφου ήδη έχουν πει πολλά. Ελέγχθη ότι η αλληλεγγύη είναι ένα σημείο κλειδί και που λείπει στην πολιτική ασύλου αυτή τη στιγμή και η απόφαση για τη μετεγκατάσταση ήταν από, από τα πρώτα βήματα για περισσότερη αλληλεγγύη στον τομέα του ασύλου. Ε, ήταν ένα βήμα όπου αποφάσισαμε επιτέλους από τους 60.000 αυτούς ανθρώπους ε, να μετακατασταθούν σε κάποια άλλα Είδαμε ότι αυτό γίνεται και ότι είναι απαραίτητη αυτή η αλληλεγγύη. Ε, απέναντι και στους πρόσφυγες, οι οποίοι φεύγουν από πολέμους, από διώξεις. Ε, ταυτόχρονα είναι έδειξε ότι μπορεί να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι λειτουργεί. Και ότι το πρόβλημα δεν είναι στις Βρυξέλλες. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν σέβονται τις υποσχέσεις τους, δεν τις τηρούν. Δεν επιδεικνύουν αυτή την αλληλεγγύη απέναντι σε άλλα κράτη-μέλη, αλλά και απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη. Αυτοί είναι σε κρίση, δεν έχουμε εμεί κρίση, αυτοί οι άνθρωποι είναι σε κρίση. Είναι σημαντικό λοιπόν το relocation είναι πολύ σημαντικό όμως ε, να εφαρμοστεί κιόλα. Βεβαίω ε, δεν είναι μακροπρόθεσμη λύση και το relocation. Υποτίθεται θα γινόταν ε, μία φορά. Πιο μακροπρόθεσμα χρειαζόμαστε μεγαλύτερου περισσότερου μηχανισμού αλληλεγγύη Είναι ένα διαφορετικό Δουβλίνο, όπω ε, ε, υπόθηκε και από την εισηγήτρια, χωρί να θίγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, χωρί να επιβαρύνονται τα κράτη-μέλη με διαδικασίε όπω αυτέ που υπάρχουν σήμερα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι μιλάμε για ανθρώπου. Οι πρόσφυγε είναι άνθρωποι έχουν οικογένεια, έχουν προτιμήσεις για το που θα πάνε, έχουν δεσμούς. Πρέπει, θέλουμε να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι και πιο εύκολο για τις χώρες υποδοχής τους να πάνε σε χώρες που θέλουν να πάνε. Δεν είναι απλά αριθμοί. Πρέπει η ένταξή τους στη συνέχεια να λειτουργήσει και να δώσουμε μια νέα προοπτική στους ανθρώπους αυτούς που έχουν φύγει από τις χώρες τους και κανείς δεν το κάνει αυτό με τη θέλησή του. Ευχαριστώ πολύ Σκά. Και τώρα ο στρατηγός ε, Άντριε Λιζιτάριου από την Ιταλία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο συνάδελφος, ο Ναύαρχος Μελώνες σας είπε ποιες ήταν ε, οι δραστηριότητες μας στην ε, Μεσόγειο. Και μέσα στο λίγο χρόνο θα ήθελα να σας μιλήσω και εγώ για τη δραστηριότητα της αστυνομίας στη Μεσόγειο. Εμείς ως αστυνομική δύναμη που δρά στη θάλασσα ε, προβάλλει διαφορετικές τεχνικές από αυτές ε, του ναυτικού και δεν έχει καμία σχέση με στρατιωτικές επιχειρήσεις. Θέλουμε λοιπόν να αναχαιτήσουμε την απειλή όταν είναι πραγματική απειλή και πρόδειλη. Γι' αυτό έχουμε το δικό μας πλαίσιο δραστηριότητας και μέσα στα πλαίσια συνεργασίας με τη Frontex δηλαδή υποστηρίζουμε τις δραστηριότητες της ε, Frontex, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης του Τρίτονα, που είναι κοινή επιχείρηση με τη Frontex. Επίσης έχουμε ε, ακτοφυλακή και δρούμε και από αέρος και από θαλάσσεις με ε, ελικόπτερα και σκάφη. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, από το 2015 μέχρι το 2017, συμμετείχαμε σε 3.000 ε, επιχειρήσεις καταστολής της παράνομης ε, μετανάστευσης και αντιμετωπίσαμε 40.000 ε, ε, διελεύσεις και φυσικά καταφέραμε να συλλάβουμε και 40 διακινητές με τα σκάφη τους. Έτσι μπορέσαμε στα πλαίσια του Τρίτονα να κατάσχουμε 9 τόνους ε, μαριχουάνας και χασίς. Όπως είπε και ο πρόεδρος Σταγιάννη σήμερα για την ανάγκη πρικοδότησης της Frontex και σε εσωτερικό επίπεδο και σε νομοθετικό και κυβερνητικό, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει κατά πιο προθυμένο τρόπο στη Μεσόγειο. Ο Κωνσταντίνος Μορφίδης τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ μέλος του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για τη σημερινή εκδήλωση. Για, για μας που αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα στην πρώτη γραμμή είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Κυρίες και κύριοι, ο ελληνικός λαός βιώνει εδώ και 7 περίπου χρόνια μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση, η οποία φτωχοποίησε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Μια κρίση που είναι παράλληλα ανθρωπιστική και κοινωνική. Όμως παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, από την πρώτη στιγμή ο ελληνικός λαός και η ελληνική πολιτεία επέδειξαν μια πρωτοφανούς ένταση και έκταση αλληλεγγύη προς τους δοκιμαζόμενους πρόσφυγες και τίμησαν τις ευρωπαϊκές και τις ανθρωπιστικές αξίες και αρχές. Το 96% όσων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν υποβάλει αίτημα χορήγηση ασύλου και βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο ικανοποίηση των αιτήσεων. Η ελληνική πολιτεία μερίμνησε για την πλήρη υγειονομική κάλυψη όλων των προσφύγων και των μεταναστών. Παράλληλα, εξασφάλισε την ένταξη των προσφυγόπουλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εμπειρία που αποκομίσαμε ω χώρα τα δύο χρόνια τη όξυνση τη προσφυγική κρίση μα επιτρέπει να βγάλουμε μερικά χρήσιμα συμπεράσματα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει όλοι μας να προνοήσουμε ώστε τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα είναι πύλη εισόδου να μην γίνουν αποθήκες ανθρώπων. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα έρχεται με το δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών μας στην έμπρακτη εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης καθώς και με συντονισμένες δράσεις σε όλα τα στάδια του ζητήματος. Από την αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης, τη μεθοδομένη και συνεχή έρευνα και διάθεση στη θάλασσα, μέχρι τη δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων υποδοχής και ένταξης. Σημαντική είναι επίσης η λειτουργία ενός δίκαιου και βιώσιμου μηχανισμού για τον αυτόματο ή σοβαρή διαμερισμό των μεταναστών και των προσφύγων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και τις προτιμήσεις των ίδιων των μεταναστών και προσφύγων. Έτσι εξασφαλίζεται η ισοκατανομή της ευθύνης μας απέναντι στους πρόσφυγες του πολίτε στον χώρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικώ έμπρακτη υλοποίηση του οράματο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση με ανθρώπινο πρόσωπο. Η συνθήκη του Δουβλίνου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη και ω εκ τούτου σε λάθο κατεύθυνση. Επομένω, θα ήταν καταστροφικό να επιμείνουμε στο λάθο και να χτίσουμε στα θεμέλια μια αποτυχημένη συνθήκη. Κυρίε και κύριοι, η Ευρώπη των αξιών και τη δημοκρατία θα πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ να σκύψει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο πρόβλημα των χωρών και των των προσφύγων. Πρέπει να μιλήσουμε επιτέλου με υπευθυνότητα για τον τερματισμό του πολέμου, για τη διασφάλιση τη ειρήνη και τη δημοκρατία και τη ευμάρεια στι χώρε που ε, δοκιμάζονται από σειράξει. Μία κουβέντα μόνο, πρέπει περισσότερο από ποτέ σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφύγει να γίνει μια μεγάλη ΜΚΟ, χωρί πολιτικέ εχμής για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματο στη ρίζα του. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σαμέρς ε, από την ομάδα του Open Delta του Μαχιλέν. δημάρχος του Μαχιλέν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Θα μιλήσω ως δήμαρχος, γιατί για έναν δήμαρχο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν είναι στατιστικά στοιχεία, είναι άνθρωποι. Είναι τμήμα των πολιτών της πόλης μας. Αυτό θέλει να είναι. Νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο μέσω στο οποίο θα μπορέσουμε να κάνουμε τη μετανάστευση κάτι επιτυχίες, ε, μια επιτυχία. Πέντε στοιχεία. υπάρχει ανάγκη να κάνουμε τα πράγματα στο σοβαρά, να καταλάβουμε ότι σε μια πολύμορφη κοινωνία υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν σαφέστεροι κανόνες και σε μια πόλη όπου υπάρχει τόση πολυμορφία θα πρέπει να κάνουμε επιπλέον προσπάθεια για να ενισχύσουμε την ελευθερία και όλων. Θα πρέπει κατά δεύτερο να δώσουμε στους μετανάστες τη δυνατότητα να αποτελούν ένα μέσο για πραγματικά προστιθέμενη άξια, να μάθουν την γλώσσα της χώρας και να είναι σαφής η εκπαίδευσή τους. Κατά τρίτον, να καταπολεμήσουμε την απομόνωση και να αποφύγουμε τον ε, στιγματισμό των ανθρώπων. Να μην θεωρούνται ούτε θύματα, ούτε εγκληματίες, ανεξάρτητα από το τι έχουν πετύχει στην προσωπική του ζωή. Να δημιουργηθεί μία κοινότητα κατά τέταρτον να χρησιμοποιήσουμε τις αξίες μας, να είμαστε σαφείς για το ποιε είναι οι αξίες μας, αλλά ποτέ ως εργαλείο αυτό για να εξαιρούμε και να απομονώνουμε άλλους, μόνο για να τους συμπεριλαμβάνουμε στους κόλπους της κοινωνίας. Και σκοπός να είναι η χειραφέτηση του καθενός. Και εδώ νομίζω ότι είναι λάθος οι λαϊκιστές. Τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω, να μην ξεχνάμε ότι ο πυρήνας της κοινωνίας μας, αυτό που την καθιστά τόσο ελκυστική, είναι ότι Υποσχόμεθα σε όλους ότι αν εργαστείτε καλά και αν ε, κάνετε ό,τι μπορείτε, μπορείτε να καλύτερε για τα παιδιά σας. Ο ρατσισμός, η διακριτική μεταχείριση καταστρέφει αυτό το όνειρο, καταστρέφει τον ιστό της κοινωνίας μας. Να καταπολεμήσουμε λοιπόν το ρατσισμό και την διακρατική μεταχείριση. Αυτό σημαίνει ότι προσπιζόμαστε την ίδια την κοινωνία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Τζόρντι Μαρτί Ντελαβούα από, την Ισπανική Γερουσία, την ομάδα Γκουε, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ε, στην Καταλωνία θεωρούμε ότι βεβαίως η κρίση των προσφύγων είναι μια παγκόσμια κρίση και βεβαίως έχει να κάνει με τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προστασίας των τροπίνων δικαιωμάτων, την πρόσπιση της ειρήνης και της ευημερίας. Στην ισπανική περίπτωση η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί ότι θα ε, υποδεχθεί 17.000 ανθρώπους και έχουν φτάσει μόλις χίλιοι. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Αφενός ένα σύστημα ασύλου το οποίο είναι προβληματικό δεν λαμβάνει, χώρα, δεν λαμβάνει υπόψη τις περιφέρειες, ε, τους δήμους, ε, τις διάφορες ε, περιοχές που θέλουν να υποδεχθούν ανθρώπους και αυτό μειώνει τη ζήτηση. Επίσης υπάρχει πολλή γραφειοκρατία, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπει να έχει κανείς πρόσβαση. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, την τοπική της Καταλωνίας, εμείς υποβάλαμε μια πρόταση για να υποδεχθούμε 4.500 ανθρώπους στην περίοδο 2015-2017. Μια πρόταση που έτυχε πολύ θετική υποδοχή από τον Επίτροπο Αβραμόπουλο αλλά και από την υποδιαρμοστία των ε, Ηνωμένων Εθνών, αλλά δυστυχώς ε, δεν οδήγησε πουθενά. Δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με την Ισπανική κυβέρνηση στον τομέα του ασύλου, διότι αυτό το σύστημα, το κεντρικό, το συγκεντρωτικό, δεν μας το επιτρέπει. Επίσης διαθέσαμε 1.200 θέσεις ε, ε, κατεπηγόντως, από τις οποίες 750 ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Τον περασμένο Φεβρουάριο περίπου 500.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Βαρκελόνης ζητώντας ε, ε, από τις αρχές ε, να αρχίσουν να υποδέχονται τους πρόσφυγες χωρίς να ψάχνουν περαιτέρω προσχήματα. Έχουμε το πρόγραμμα Καταλωνία για τους πρόσφυγες έτσι ώστε αυτό το σύστημα του Ισπανικού κράτους που οδηγεί στο ότι πολλοί άνθρωποι μένουν εκτός της κάλυψης να μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε με τη βοήθεια, της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό που ζητάμε εμείς ως Ρεπουμπλικανική Αριστερά της Καταλωνίας ε, να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι στην Καταλωνία. Ευχαριστώ από την Πολωνία τώρα. Ε, Επιτροπή των Περιφερειών έχει κάνει τη γνωμοδότηση για την παράνομη μετανάστευση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια από την ε, Επιτροπή των ε, Περιφερειών σε σχέση με την ε, μετανάστευση. Συμφωνώ απόλυτα με τον Επίτροπο, ο οποίος τόνισε ότι εάν θέλουμε να σταματήσουμε την παράνομη μετανάστευση θα πρέπει να ανοίξουμε νόμιμους διάβλους στην Ευρώπη, γιατί όταν μιλάμε για παράνομη μετανάστευση, μιλάμε για το μέλλον μας, για το μέλλον της Ευρώπης, για την ανάπτυξή της και για το μέλλον της Ευρώπης που αναπτύσσεται για τα παιδιά μας. Και αν θέλουμε καλύτερη ανάπτυξη θα πρέπει να έχουμε ανθρώπους που προέρχονται από ολόκληρο τον κόσμο γιατί υπάρχουν πολλές ελλείψεις στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το δημογραφικό πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε τη μεταρρύθμιση της μπλε κάρτας, έτσι ώστε να ε, μπορέσουν να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι και στις δικές μας χώρες. Επίσης, θα πρέπει να τονίσω ότι εκπρόσωπος από τα Ηνωμένα Έθνη προηγουμένως τόνισε ότι θα μπορούσαμε να δράσουμε πιο στοχοθετημένα ιδιαίτερα από πλευράς χωρών όπου δεν υπάρχουν ε, μετανάστες, δεν υπάρχουν πρόσφυγες, με συγχωρείτε φαίνεται ότι ισχύει μια κατάσταση σαν να πρόκειται για ένα φόβητρο. Όμως και στην Πολωνία θέλουμε να καταδείξουμε την αλληλεγγύη μας, αλλά θέλουμε ειδικά προγράμματα ε, έτσι ώστε να προωθήσουμε τη συνεργασία με τους περιφερειακούς φορείς. Ο, ο Δήμαρχος της Κατάνια έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από τρεις μήνες στην πόλη μου, την Κατάνια, στο λιμάνι, είχαμε ένα στρατιωτικό σκάφος, Έιτνε ονομάζεται, και επεβιβάζονταν 700 άτομα. Το σκάφος αυτό αυτό ήταν ε, μια ακόμα περίπτωση. 716 ήταν τα άτομα τελικά, διότι γεννήθηκε εμπλό ένα μωρό ε, του οποίου ε, επέζησε η μητέρα αλλά όχι ο πατέρας. Χάθηκε ενώ άλλαζαν σκάφη κατά το ταξίδι τους στη θάλασσα της Εκελίας. Στην πόλη με αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από χίλιοι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Το 2016 στις ακτές της Ικελίας έφτασαν 200.000 άτομα. Μόνο στην πόλη της Κατάνια 20.000 περίπου. Από αυτούς είναι μεγάλος αριθμός των ανηλίκων και έχουν φτάσει και σωροί, τους οποίες ε, έχουμε θάψει στο νεκροταφείο. 221 ε, σωροί στο νεκροταφείο της ε, Κατάνια. Ένας νεαρός Σύριος, Σύρος συγκεκριμένα, ο οποίος τραυματίστηκε σε βομβαρδισμό ε, σε βομβαρδισμούς σε πόλη της Συρίας, ε, δέχτηκε περίθαλψη στην Φλωρεντία και τελικά κατέληξε στην πόλη μου. Έχουμε αισθανθεί εγκαταλειμμένοι, ε, Πρόεδρε, πολύ μόνοι τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πολλές φορές την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταλάβει το πόσο σοβαρό είναι το φαινόμενο. Για μας σήμερα η μέρα είναι πολύ σημαντική. Ε, συμφωνώ απολύτω, με τις προτάσεις που άκουσα από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Ευρωπαίο Επίτροπο. Ζητούμε το δικαίωμα στο άσυλο να ε, θεμελιώνεται σε ευρωπαϊκά ε, κείμενα. Δεν γίνεται να έρχονται άνθρωποι από τη Συρία και να θεωρείται ότι μπορεί να μην έχουν δικαίωμα να αιτηθούν άσυλο. Πρέπει να είναι μια ευθύνη κοινή η διαχείριση των προσφύγων. Πρέπει οι τοπικέ κοινότητε ε, να ενισχυθούν στην προσπάθεια να βοηθήσουν του πρόσφυγε. Και για την νομοθεσία ε, καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων που οργανώνουν την εμπορία ανθρώπων. Πρέπει κάτι να γίνει όπω και για την πολιτική στήριξη τη Λιβύη. Σα ευχαριστούμε για αυτέ τι πρωτοβουλίε. Πρόεδρε, αισθανόμαστε κάπω λιγότερο μόνοι. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετική η μαρτυρία σας, συνάδελφοι. Μου λένε ότι έχουμε ακόμα 20 λεπτά. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πότε θα τελειώσει αυτό το πάνελ. Διότι έχουμε ακόμη 15 ομιλητέ. Ποτέ δεν είχα ένα κατάλογο τόσο μακροσκελή όλη μου την ε, ζωή. Και δεν ξέρω και τι θα κάνω, αλλά η διαφορά εδώ είναι ότι έχουμε τέτοιε παρεμβάσει όπω η τελευταία που είναι πραγματικά κέρυε. Είναι σοβαρότατε. Δεν μπορούμε να διακόψουμε τη συζήτηση. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που έχουν να πούν όλοι και πρέπει όλοι να πάρουν το λόγο. Ε, όλοι έχουν παραμείνει περίπου στα δύο λεπτά. Δεν είναι λοιπόν ότι κάποιο είναι πιο πειθαρχημένο από τον άλλο. Ε, ούτε είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αρχίσαμε με μια ώρα καθυστέρηση. Προτείνω για τους 15 αυτούς ομιλητές να παραμείνουμε σε περίπου ένα λεπτάκι. Θα με διευκολύνατε πάρα πολύ. γιατί έτσι θα παραμείνω στο τέλο αυτού του πάνελ, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν μπορώ να σα κόβω. Παρακαλώ να προσπαθήσετε να είστε σύντομοι. Ο κ. Κάλκαν, γραμματέα τη ε, Επιτροπή Δημάρχων, για δύο λεπτά. Εάν μπορέσετε και σένα, βέβαια, καλύτερα ακόμα. Η κυρία Κάλκαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω εκ μέρου τη Επιτροπή των Δημάρχων. Είμαστε μια ανεξάρτητη ε, οργάνωση από τι κάτω χώρε και αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην καρδιά τη μεταναστευτική πολιτική να υπάρχει εξωτερική ύψη τη πολιτική ασύλου και μετανάστευση. Το βλέπουμε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όπω πρόσφατα στην Ολλανδία. Επίση, ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει την τέταρτη έκθεση προόδου για τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει τη Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη μετανάστευση. Ε, παρόλο που τα μέτρα και τα στοιχεία που έχουμε είναι θετικά σχετικά, ε, βλέπουμε ότι δεν έχουν ε, πλήρως τα περισσότερα κατεμέρια της του υποχρεώση, υποχρεώσεις, ιδίως ό,τι αφορά το σύστημα τη επανακατάστασης. τη μετακατάσταση, μάλλον. Το, η πρόοδος είναι πολύ βραβεία και οι περισσότεροι δεν έχουν κάνει τίποτα. Ε, παρόλο που κάποιοι το, το παρουσιάζουν το σύστημα αυτό ω επιτυχημένο και παρά τι επικρίσει τη κοινωνία των πολιτών και των ακαδημαϊκών, ε, των πανεπιστημιακή κοινότητα. Η Τουρκία ε, σύναψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να ασφαλή ούτε χώρα όπου ήταν βέβαιο το ότι θα αποκίνουν οι πρόσφυγε. Το σύστημα ασύλου λοιπόν απαιτεί θεμελιώδει επιλογέ για την ε, ε, επανακατάσταση και την επιστροφή. Θα πρέπει το σύστημα αυτό να είναι ευρωστό, να είναι ανεξάρτητο και να λαμβάνονται αποφάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σοβαρά για το θα υπάρχει συνεργασία με τρίτε χώρε. Η μόνη Αφρικανική χώρα που βάσει αντικειμενικών πληροφοριών είναι ασφαλή για του πρόσφυγε είναι το Μαρόκο. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε σε κριτήρια που θα συμφωνηθούν μεταξύ των κρατών ε, μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να βρούμε και άλλα κράτη εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι πρόθυμα να συνεργαστούν. Ε, δεν τα καταφέρνω σε ένα λεπτό, ε, όσο και αν είμαι σύντομη. Θα πρέπει επίση να δούμε τι ε, ε, ακούστηκε στην διάσκεψη που έγινε στι 18 Μαου στη Χάγη και για να συνοψίσω υποχρεώσει των κρατών μελών βάσει του διεθνού δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου ε, είναι να ε, παρακολουθούνται και να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν συμφωνίε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτων κρατών για να διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ετών άσυλων, των προσφύγων, των μεταναστών και πάντα τα βρίσκεται και στον τοπό μα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από το Φλαμανδικό ε, Κοινοβούλιο, από, την, από το κόμμα NVA, για ένα έω δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όντως μιλώ ως μέλος της ε, Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά και ως μέλο του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου εδώ στις Βρυξέλλες. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όμως το κλειδί τη στρατηγικής είναι η ένταξη. Η ένταξη και η συνοχή σε τοπικό επίπεδο που πρέπει να ενισχυθεί. Θα πρέπει να εντάξουμε τους νέου ερθέντε της κοινωνία μας. Θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος της κοινωνίας μα. Ε, δεν πρέπει δηλαδή να θεωρούνται παρήσακτοι η έκθεση για την ένταξη στην Επιτροπή μας που βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές ε, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις βέλτιστες πρακτικές ε, της φλαμανδικές εδώ και χρόνια. Η Φλάνδρα κάνει μια προσπάθεια ε, για μια πολιτική ένταξη που βασίζεται σε δύο αρχές. Πρώτα να μάθουν οι άνθρωποι τη γλώσσα. Αυτό τους επιτρέπει να μπορούν να έχουν μια διάδραση με το περιβάλλον τους η δεύτερη αρχή είναι ε, η, η ένταξη ως πολίτες στην κοινωνία. Ε, όχι μόνο ε, επειδή τους δίνουμε χαρτιά, αλλά και στο κεφάλι τους και στην ψυχή τους. Ε, αυτό θα μας βοηθήσει να οργανώσουμε καλύτερα την κοινωνία μας, να καταλάβουν και αυτοί καλύτερα πώς λειτουργεί το κράτος δικαίου, η δημοκρατία οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι οι πρώτες οντότητες που αντιμετωπίζουν την πρόκληση της ένταξης. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστώ ο Τίμπορ Βάνα, αντιπρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το κόμμα Γιόμπικ. Ένα με δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό υπό μεταναστευτικές πιέσεις υπάρχουν μεγάλη κίνδυνοι για την ασφάλεια. Πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε τις ροές αυτές για να αποτρέψουμε τις ενδυνάμει τρομοκρατικές πράξεις διότι ε, αυτό υπονομεύει και την ανάγκη διεθνού προστασίας. Η ριζοσπαστικοποίηση δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών είναι ένα άλλο πρόβλημα στις δυτικέ χώρε. Πρέπει όλε οι χώρε τη Ένωση να κάνουν ό,τι μπορεί να προστατεύσουν τα σύνορά του. Στην Ουγγαρία άρχισε να φτιάχνει το φράχτη στα σύνορά τη για να προστατεύσει το έδαφο τη Σέγγεν πιο αποτελεσματικά. όλε οι άλλε χώρε μα κατηγόρησαν για παραβίαση των δικαιωμάτων. Τώρα όμω ε, η προστασία των εξωτερικών συνόρων έχει γίνει προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι τώρα είναι σαφέ ότι η Ουγγαρία έκανε τη σωστή, ε, πήρε σωστή απόφαση, έκανε σωστή επιλογή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να επιληθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν κάνουμε σημαντικά βήματα στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες, αυτή η ροή δεν θα σταματήσει και η Ευρώπη που γνωρίζουμε τώρα θα αλλάξει για πάντα. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά τις χώρες εκείνες που πρέπει να προστατεύσουν τα σύνορα Σέγγεν. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ από το Μεσογειακό Παρατηρητήριο Μετανάστευσης ε, Προστασίας και Ασύλου για λιγότερο από δύο λεπτά παρακαλώ. Είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Middlesex και ε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι ένα ειδικό σχέδιο για τη μετανάστευση. Αυτό έχει μεγάλη σημασία η αντιμετώπιση των ε, μεταναστών από πλευράς φύλου, ηλικία και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές για την αντιμετώπιση των μεταναστών που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Και επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το καθεστώς χορήγησης ασύλου σε αυτούς που το χρειάζονται. Να δούμε τους, ε, τις ευάλωτες κατηγορίες, ιδιαίτερα αυτούς με νοητική υστέρηση. Στο ε, ε, Coventry, Warwick και άλλα πανεπιστήμια τονίσαμε στις μελέτες ότι θα πρέπει να υπάρχει ασφαλής μετάβαση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ξέφυγαν από τον πόλεμο, το λοιμό και τη, τη δολοφονία. Δεν ε, δεχόμαστε τα απάνθρωπα ε, στην ουσία σαν στρατόπεδα κράτησης, ε, γιατί δεν πρόκειται για πραγματικά καταλήματα. Ειδικά από πλευράς Νορβηγίας και Φιλανδίας, όπου δυστυχώς υπάρχουν απάνθρωπες ε, συνθήκες κράτησης. Είχαμε ε, έναν ε, πρόσφυγα ο οποίος έκανε απεργία πείνας για 65 μέρες και θυματοποιήθηκε από την ε, αστυνομία. Αυτός ε, ο πρόσφυγας βρίσκεται τώρα στην Αθήνα. Ε, Μαρία Μποργέζιο από την ομάδα ΙΕΝΕΦ για ένα με δύο λεπτά. Έχουμε να κάνουμε με μία κατάσταση κατάσταση πολιορκίας και κανένας δεν έκανε τόση σχετισμό μεταξύ ε, μετανάστευσης και τρομοκρατίας. Γιατί οι τρομοκρατικές οργανώσεις βασίζονται στους παράνομους μετανάστες. Έχει μεγάλη σημασία ο επαναπατρισμός των ε, μεταναστών, ιδιαίτερα στους 18.500 ε, Νιγηρινούς που έφτασαν στην Ιταλία, μόνο το 3% ε, έχει το δικαίωμα να παραμείνει. Οι άλλοι που βρίσκονται παραμένουν δυστυχώς στην Ιταλία ή μεταβαίνουν το πολύ στη Γαλλία. Κανένας δεν τους διώχνει από τη χώρα. Μόνο 120 εκδιώχθηκαν. Γι' αυτό ε, μία συγκεκριμένη ΜΚΟ είχε μία περίεργη δραστηριότητα. Όπως ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο της προστασίας των θαλασσίων σύνορων. Έγινε μία εξεταστική επιτροπή η οποία ασχολείται με το σύνδεσμο αυτών των ΜΚΟ και των διακινητών. Και γι' αυτό θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή τη ε, διακίνηση. κυρία Μοκερίνη είναι πολύ υπερήφανη για τα αποτελέσματα, μα είναι υπερήφανη και για τον τρόπο υποδοχής των μεταναστών από τη Συρία που δίνουμε από την Ευρώπη που όλο υποκρίνεται στον κύριο Ερντογάν και σε αυτό το ερώτημα θα έπρεπε να ε, απαντήσουμε. Hans Gustav Mersberg από το ε, ελεγκτικό συνέδριο. Ένα με δύο λεπτά θα ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα των hot spots από πλευράς ελεγκτικού συνεδρίου. Μας ενδιαφέρει να δούμε κατά πόσο έχουν συσταθεί εγκαίρως και κατά πόσο η προσέγγιση ήταν αποτελεσματική έτσι ώστε να έχουμε πλήρη ε, αναγνώριση, καταγραφή και δακτυλοσκόπηση των ε, μεταναστών και τη σωστή διαχείριση της μετανάστευσης. Δυστυχώς ήταν μια σχηνοτενής διαδικασία και δεν απαντήσαμε άμεσα σε μια κατάσταση η οποία μετατρεπόταν σε ανθρωπιστική καταστροφή. Πολλά, πολύ περισσότερα θα πρέπει να γίνουν και έχουμε και πολλές συστάσεις. Θα πρέπει να δούμε τις ανεπάρκειες των hotspot, δηλαδή αναβάθμιση των υποδομών. Όλοι οι φορείς θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουν σωστά το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων και θα πρέπει να υπάρχει υπηρεσία προστασίας των ανηλίκων, ειδική υπηρεσία για την προστασία και την κυδαιμονία τους και η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει την πραγματογνωμοσύνη για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την εξωτερική μαρτυρία. Ο κύριος Ιγνάσιο Γκαρθία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τους Μετανάστες στην Ευρώπη. Καλησπέρα σας, Πρόεδρε. Πολύ ευγενική πρόσκλησή σας σήμερα το απόγευμα. Ένα λεπτό θα προσπαθήσω. Ε, πρώτο μήνυμα. Πρέπει να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Είναι αδύνατο να λάβουμε εμείς αποφάσεις στη θέση των ε, προσφύγων για το που θα πάνε Είναι σημαντικό αυτό. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς για τους ζωές Δεύτερον, πρέπει να είμαστε πολύ πιο δημιουργικοί με την ε, ε κράτηση. Η κράτηση είναι πηγή πόνου, καταστρέφει τις ζωές των ανθρώπων και των οικογενειών. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πιο επινοητικοί και να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις. Και τρίτον, και αυτό είναι απλώς ένα μήνυμα που πρέπει να ακουστεί χειρά σήμερα το απόγευμα, εργαζόμαστε με τους πρόσφυγες αλλά και με εθελοντές, εκατοντάδες γυναίκες και άντρες σε όλη την Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ποιοι έχουν τις περισσότερες ανάγκες λοιπόν. Η κοινωνία των πολιτών έχει εργαστεί για την ε, φιλοξενία και για να υποδεχτεί τους πρόσφυγες, προσπαθώντας ε, να προστατεύσει αυτούς που έχουν ε, μπει στο περιθώριο. Πρέπει να δράσουν οι πολίτες. Φυσικά δεν περιμένουμε ε, από τους πολιτικούς ηγέτες λιγότερη αποφασιστικότητα από ό,τι έχουν δείξει οι ίδιοι οι πολίτες μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Μου φαίνεται δύσκολο να δίνω στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Συνοροφυλακής και Εκτοφυλακής μόνο ένα λεπτό, αλλά αν μπορείτε να πείτε τα βασικά σας μηνύματα σε ένα λεπτό θα σας ήμουν ευγνώμων. Έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές, οπότε ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε για την πρόσκληση, ε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Οι προηγούμενοι ομιλητέ μίλησαν για την περιπλοκότητα του φαινομένου τη μετανάστευση. Θέλω να πω ότι η διαχείριση των συνόρων είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο, ε, ξεπερνά τα όρια τη μετανάστευση και η διαχείριση τη μετανάστευση είναι ευρύτερη από τη διαχείριση των συνόρων. Η δική μα συνεισφορά ω Ευρωπαϊκή Συνοροφυλακή και Εκτοφυλακή ε, ω προ τη διαχείριση των σύνορων έχει να κάνει με την εποπτεία των σύνορων, τι περιπτώσει βοήθεια και διάσωση. Έχουμε σώσει 90.000 ζωέ μόλι πέρσι και συμβάλλουμε και στην καταγραφή των μεταναστών, ε, την ε, λήψη δακτυλοκεντρών αποτιμάτων, του ελέγχου ασφάλεια και τι επιστροφέ. Οι επιστροφέ έχουν εντατικοποιηθεί προκειμένου να έχουμε πραγματικές επιστροφές αλλά με τη σωστή ταυτοποίηση προηγουμένως αυτό είναι το καθοριστικό στοιχείο. Έχουμε επίση μια νέα εντολή ε, προσπαθώντα να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δράση. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση δυνατοτήτων εντό των κρατών μελών, αλλά και στι τρίτε χώρε. Και έχουμε και τη δυνατότητα να πετύχουμε το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ εσωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργασία με τρίτε χώρε. Όπω αυτή τη στιγμή η αποστολή εξωματικών συνδέσμων στην ε, Νιγηρία, την Τουρκία και στα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλώς το βήμα των Ευρωπαίων Νομοθετών ε, πέρσι για την αύξηση των πόρων που προβλέπονται για την Ευρωπαϊκή Συνοφυλακή και Εκοφυλακή μπορεί να φέρει μεγάλη διαφορά. Και ελπίζουμε ότι θα συνεισφέρουμε σε καλύτερη διαχείριση της νόμου μετανάστευσης καθώς και σε καλύτερη μεταχείριση, ε, προστασία μάλλον των εξωτερικών μας συνόρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε που σεβαστήκατε και το χρόνο ομιλία Και τώρα από τη Φιλανδική Βουλή των μέλος των Πρασίνων, Ευχαριστώ. Γεια σας από τη Φιλανδία. Εμείς καλωσορίζουμε το νέο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Είναι απαραίτητο. Οι συζητήσεις στη Φιλανδία ε, αφορούν κυρίως κατά πόσο αυτές οι πολιτικές πρέπει να είναι θελοντικές ή δεσμευτικές. Εγώ είμαι στην αντιπολίτευση και πιστεύω ότι οι δεσμευτικές πολιτικές είναι απαραίτητες σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να μοιραστούμε το βάρος, οι χώρες που πιέζονται πρέπει να βοηθούνται. χρειάζεται κοινό έλεγχο στα σύνορα, η εσωτερική, ε, το εσωτερικό relocation ε, είναι μια καλή λύση, αλλά πρέπει να το επεκτείνουμε περιττέρω. Εμείς αναλάβαμε το μέρος μας αναλόγως, πρέπει να το κάνουν και οι άλλοι όμως. Και αυτοί που ε, λαμβάνουν το άσυλο πρέπει να βοηθούν στη συνέχεια και να, για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους όσο γίνεται πιο ανθρώπινα. Και για όσους δεν λάβουν το άσυλο θα πρέπει να επικοινωθούμε στα μαλακά μέτρα. Ορισμένες φορές βεβαίως χρειάζονται και οι απελάσεις. Ε, και υπάρχει και το θέμα των ανθρώπων χωρί χατιά. Εκεί χρειαζόμαστε κοινέ λύσει. Είναι δύσκολο να μείνει κάποιο στη χώρα μα χωρί χατιά, λόγω και του κλίματο, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Είναι σε ευάλωτη κατάσταση αυτοί οι άνθρωποι και είναι ευάλωτοι απέναντι σε πολλέ μορφέ εγκληματικότητα. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ στο γεγονό ότι χρειάζονται ε, κοινέ ε, ευρωπαϊκέ πολιτικέ ε, οικογενειακή επανένωση. Ευχαριστώ πολύ. Μπραντου ο οποίο είναι ευρωβουλευτής του S&D στην, ε, ε, και είχε αναλάβει την έκθεση για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωκοινοβούλιο ασχολείται με την μεταρρύθμιση τη πολιτική μετανάστευση και ασύλου σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Σήμερα όμω πρέπει να θέσουμε μια προτεραιότητα με σαφήνεια. Μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, που να βάζει τέρμα στην αρχή τη χώρα προέλευση και να ορίζει ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την εξέταση μια αίτηση ασύλου. Δεν είναι μόνο μια διοικητική υποχρέωση. Ένα σύστημα που βλάπτει τα άτομα τα οποία αναζητούν ε, προστασία και ποινικοποιεί τι χώρε που βρίσκονται βρίσκονται στα σύνορα και στο πρώτο γραμμή τη μάχη, όπω η Ελλάδα και η Ιταλία. Θα πρέπει να υπάρχει συγκατανομή των ευθυνών ε, μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ξεκινούμε από αυτό το κομπικό σημείο, δηλαδή την πλήρη υλοποίηση των προγραμμάτων ε, μετεγκατάσταση. Γιατί είναι σαφέ ότι όλα αυτά σχετίζονται με την πραγματική δυνατότητα των διοικητικών αρχών να προσφέρουν όρου υποδοχή και προοπτικέ εγκατάσταση βάσει των θεμελιωτών δικαιωμάτων και τι αρχέ του διεθνού δικαίου. Δεν μπορεί να αμφιλητούνται αυτά και πρέπει να είναι βιώσιμε οι λύσει και για τι κοινωνίε που υποδέχονται του μετα... Εγώ ήμουν εισηγητή για την ε, επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των προσφυγών στα πλαίσια τη Επιτροπή Απασχόλησης στη δουλειά μου. Υπογράμμισε ένα στοιχείο πολύ σημαντικό αλλά και κέρια σημασία, δηλαδή ότι η πρόκληση τη ένταξη μπορεί να γίνει μια μεγάλη ευκαιρία αν δείξουμε ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, που ούτως ή άλλω ε, ε, καλούνται να λύσουν οι κοινωνίε μα με έναν τρόπο καθολικό, ε, σφαιρικό θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις οικογένειε των ανέργων και τι οικογένειε με χαμηλά εισοδήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Από την Ιταλική Γερουσία, ο κύριος Μάριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ λίγα λόγια, γιατί είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Για να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να δώσει μια ευρωπαϊκή διάσταση στο θέμα και μας δίνει μια μεθοδολογία για να μπούμε στην ουσία ενός ζητήματος που θα μας συνοδεύει για αρκετά χρόνια. Εγώ αναφέρομαι σε γεγονότα μόνο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για να μπορέσουμε να εργαστούμε. Η Ιταλία είναι η μόνη χώρα που έχει διπλωματική παρουσία στη Λιβύη. Στην Τίνιδα βρίσκεται το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και γραφείο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το λέω προς την ε, κυρία Μογκερίνη. Θα πρέπει να φανούμε θαραλέοι αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, φτα... Φτάσαμε σε μια συμφωνία με την Τουρκία, την Τινησία και την Αίγυπτο. Ας προωθήσουμε αυτή τη συμφωνία με σημεία αναφοράς και hot spot σε χώρες που είναι πιο ασφαλείς από τη Λιβύη και ίσως δεν είναι λιγότερο ασφαλής από την Τουρκία. Εμείς δαπανούμε δέκα δις κάθε χρόνο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα δεν μας φοβίζει η δαπάνη, αλλά το γεγονός ότι προβάλλουμε μία, προβάλλουμε μία οικονομική αντιμετώπιση η οποία μας οδηγεί πιο μακριά από τους στόχους της υποδοχής. Και άμα χάσουμε την συνένεση των Ευρωπαίων πολιτών τότε το έργο μας θα, είναι, θα γίνει ακόμα πιο άχαρο. Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος για ένα λεπτό. Ε, θα μιλήσω εκ μέρους των τοπικών αρχών. Χρειαζόμαστε ένα βιώσιμο σύστημα διαχείρισης μετανάστευσης και δεν μπορούμε πλέον απλά να αντιδρούμε στις πραγματικές κινήσεις με ανάλογα με τις εξελίξεις που βρίσκουμε. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία για την ορθή και ουσιαστική μεταρρύθμιση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου όσο το δυνατόν συντομότερα. Καλό θα ήταν το καινούριο σύστημα να λαμβάνει υπόψη τι δυνατότητε υποδοχή των μεταναστών του κάθε κράτου μέλου. Η μετεγκατάσταση των ετούντων για άσυλο πρέπει να προχωρήσει με πολύ πιο γρήγορου ρυθμού από ό,τι μέχρι τώρα. Και τέλο, η Επιτροπή των Περιφερειών έχει ζητήσει επανειλημμένα διευκόλυνση τη παροχή κονδυλίων στι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ για τη διαχείριση τη μετανάστευση. Οι πόλει στα χωριά και οι περιφέρειε, ειδικά κοντά στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, υφίστανται μεγάλη πίεση και συχνά δεν έχουν τα μέσα να την αντιμετωπίσουν. Πρέπει επίση να σα πω ότι όλε οι πολιτικέ παρατάξει τη Επιτροπή των Περιφερειών συμφωνούν με τον κύριο Ταγιάννη, με τον κύριο Γιούγκερ και βεβαίω με τον Κομισάριο τον κύριο Αβραμόπουλο. Για πρώτη φορά βλέπουμε ότι ακούγονται, γιατί πολλέ φορέ η Ευρώπη ασχολείται με μεγάλα κάνει μεγάλα πράγματα, παραδείγματο χάρη τη διατήρηση του γάλα του 7 ημερών και άλλα θέματα τα κάνει πολύ, πάρα πολύ μικρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σκύβεται στο θέμα. Είναι τεράστιο, εξαρτάται το μέλλον τη Ευρώπη. Δεν θέλω να μιλήσω για την Ελλάδα, είναι γνωστό σε όλου τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σα ευχαριστώ και τελευταίο ο ε, Δεν ε, το πίστευα, αλλά φτάσαμε στο τελευταίο. Τουλ, πρόεδρο του Royal Europa ε, Initiative το ενοποίηση μέσω του αθλητισμού. Έχετε λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να ολοκληρώσω τις παρεμβάσεις. Είμαι ο επικεφαλής ε, του μια λέξη και στο Κράινεμ, όπου πριν από δύο χρόνια αποφασίσαμε να καλωσορίσουμε ε, νέους, νεαρούς, ασυνόδευτους ε, πρόσφυγες. Κάθε μέρα έρχονται Έξι έως 10 νεαροί πρόσφυγες, με τους οποίους μαθαίνουμε γαλλικά ή ολλανδικά. Κάνουμε παιχνίδια, αθλητικά και... Πρόκειται για άτομα που έρχονται από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ, από χώρες που υπάρχει πόλεμος και η μοναδική τους ελπίδα είναι να μπορέσουν να ενσωματωθούν με επιτυχία. Αυτό για να σας υπογραμμίσω τη σημασία του αθλητισμού ως παράγοντα ενσωμάτωσης. Χρειάζονται πολύ ε, πάθος, θέλοντες, ε, θέληση για να το πετύχουμε αυτό και πολλή δουλειά. Υπάρχει μια πολυπολιτισμική πλατφόρμα άτομα από 350 διαφορετικές οικογένειες. Πάρτε λοιπόν το κινητό σας ε, πάρτε την κατεύθυνση του αεροδρομίου και σταματήστε στο Κράινεμ να δείτε αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία για τους νεαρούς πρόσφυγες. Σας ευχαριστώ. Είναι πραγματικά αισιόδοξη η νότα αυτή κλείνοντας. Δεν πρόκειται να κάνω μεγάλη καταληκτική ομιλία γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει 50 λεπτά. Ζητώ συγγνώμη στην επόμενη, από την επόμενη, τους οργανωτές της επόμενης συνεδρίασης. Δεν φταίγαμε εμείς όμως να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μίλησαν τα τελευταίοι που έδειξαν τόσο μεγάλη υπομονή και επιθερχία. Νομίζω ότι είχαμε 40 ομιλητές και θα σας αναφέρουμε και θα ανακεφαλαιώσουμε τις εξαιρετικές αυτές παρεμβάσεις στην τελική συνεδρίαση. Και τώρα να δώσουμε το λόγο για τον τρίτο γεωτραπέζι, για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Αγκουστίν Διασδεμέρα θα είναι ο πρόεδρος της τελευταίας αυτής ε, συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ πολύ.